Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. L'ordre du jour. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε βεβαρημένη μερισιά διάταξη. La séance est ouverte. Κήρυξω την έναρξη της συνεδρίασης. Μία σειρά συνεδριάζουν βέβαια, διότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί και αύριο το απόγευμα. Θα ήθελα να σας πω ότι από ό,τι φαίνεται, αύριο το πρωί θα είχαμε μία μακρά ανταλλαγή απόψεων για την εξέταση των οργανισμών, 9 με 11 θα γινόταν αυτή η ετήσια συνεδρίαση, ε, μάλλον η ανταλλαγή απόψεων, ε, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα στις 10, μέχρι τις 10 να το έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα. Επομένως, λέω, αντί να ξεκινήσουμε στις 9, να ξεκινήσουμε στις 9 και μισή αύριο. συμφωνείτε με το σχέδιο μέσιας διάταξης. Ο κύριος Ντεπρέ, από ό,τι βλέπω, θα ήθελε το θέμα που πρόκειται να συζητηθεί σήμερα υπό το 8 σύστημα πληροφοριών και άδεια ταξιδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΤΙΑΣ. Δεν μπορεί ο κύριος Ντεπρέ να είναι απόψε εδώ. Θα ήθελε λοιπόν να το δούμε το θέμα αυτό αύριο μεταξύ 10 και μισή και 11 παρα 10. Με αυτή την τροποποίηση και αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκρίνεται με τις δύο τροποποίησεις που προανέφερα η μερίσια διάταξη. Η διαπραγματευτική ομάδα της ε, Επιτροπής μας υπό την Έντερ Γκουαρδιαθάμπαλ για δύο νομοθετικά ζητήματα που εντάσσονται στο, εξωτερικό, στο σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων, βιώσιμες επενδύσεις και την εξωτερική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Εξωτερικές Δράσεις Μέχρι στιγμής δεν κατέληξε σε συμφωνία στον τρεμερή διάλογο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε οι διαπραγματεύσεις ε, θα επαναληφθούν μετά τις θερινές διακοπές και θα κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης αυτής ε, στην προσεχή μας συνεδρίαση. Και αυτό παρά τις προσπάθειες ε, που έχει καταβάλει η ΕΝΤΕΡ, που πραγματικά ήταν επίπονες οι διαπραγματεύσεις αυτές και οι δικές προσπάθειες Μεγάλης. Αυτά είχα να πω, αυτές ήταν ανακοινώσεις και ερχόμαστε στο εργαστήριό μας που αφορά τις διαδικασίες για τον προϋπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι ένα εργαστήριο προβληματισμού το οποίο διοργανώνεται κατόπιν ετήματος των μελών της Επιτροπής Μπάτζ και στόχο έχει να δοθούν πιο πολλές πληροφορίες για την λειτουργία ε, του γεωργικού προϋπολογισμού υπό την κατηγορία 2 του ετήσιου προπολογισμού και ιδίως ό,τι αφορά τη διορθωτική επιστολή για το σχέδιο προπολογισμού στον τομέα της γεωργίας. Εγκρίνεται κάθε Σεπτέμβριο Κάθε δηλαδή φορά έχουμε το Σεπτέμβριο μία διορθωτική επιστολή. Εμείς αποφασίσαμε το εργαστήριο να το οργανώσουμε πριν το καλοκαίρι για να δοθεί δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής μας να λάβουν πληροφορίες που θα τους είναι απαραίτητε για το θέμα αυτό πριν λήξει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τον προβλησμό 31 Αυγούστου λίγη πλέον φέτος αυτή η προθεσμία. Τα χαρακτηριστικά του γεωργικού προβλησμού είναι ότι ξεκινάει 15 Οκτωβρίου το έτος, αν θέλετε, και ολοκληρώνεται, όχι, 16 Οκτωβρίου στη χρονιά νη, νημιονένα και λίγη στις 15 Οκτωβρίου της χρονιάς νη. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της γεωργίας, για να γίνουν και απαραίτητες προσαρμογές όταν έρχεται η ώρα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και λαμβάνουμε, όπως είπα, κάθε χρόνο μια διορθωτική επιστολή λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, προβλέψεις ε, και τις ε, συστάσεις του Κοινοβουλίου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκέοργ Χόισλερ, που είναι ο Διευθυντής Πόρων της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Γεωργία Ανάπτυξης Πέτρο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήρθε εδώ για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την όλη αυτή διαδικασία, την ετήσια διαδικασία του προπολογισμού. Πριν δώσω το λόγο στον προσκεκλημένο που θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ σήμερα, Θα ήταν καλό σας να ακούσουμε καταρχάς τους δύο μόνιμους εισηγητές για τον γεωργικό προϋπολογισμό. Άσχουερτ και Αλή. Ο κύριο Αλή δεν είναι εδώ όμως. Παρ' όλα αυτά μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα προβληματισμού που αφορά πιο πολύ το περιεχόμενο και όχι τόσο τη διαδικασία που η παρουσίαση αφορά πιο πολύ την, παρουσία, την διαδικασία, τη μεθοδολογία δηλαδή και όχι το περιεχόμενο του γεωργικού προπολογισμού. Θα σας δώσω ένα αντίτυπο αυτού του σημειώματος ώστε και εσείς ε, να ενημερωθείτε για τις παρατηρήσεις του. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνεισηγητή, τον κύριο Ρίζαρ Ντάσκοτ. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ε, Γεωργίας και πώς λειτουργεί στον τομέα αυτό η όλη διαδικασία. Συνάδελφοι, ζήτησα να γίνει η συζήτηση αυτή, γιατί είναι τεράστιο όγκο τεχνικών λεπτομεριών που συχνά δεν γίνονται κατανοητέ. Και γι' αυτό καλωσορίζουμε τον Γιώργο Χόισλε που είναι εδώ σήμερα για να μα βοηθήσει να τα καταλάβουμε καλύτερα. Πιο συγκεκριμένα, θα ενδιαφέρει το θέμα του συναδέλφου, γιατί πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα πώς το σύστημα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί μπορούν να ανταποκριθούν σε προβλήματα που επηρεάζουν την όλη βιομηχανία. Εάν δούμε αυτή την περίοδο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, είχαμε δυσκολίες όπως έκτακτες περιπτώσεις, όπως το εμπάργκο στο ρωσικό εμπόριο. Ε, την, τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά και τις αλλαγές των ισοτιμιών. Αυτά πιέζουν το ε, εισόδημα και πρέπει οι μηχανισμοί χρηματοδότησης να δείξουν την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμοστούν. για να βρεθούν οι κατάλληλε λύσει για τι εταιρείε του χώρου. Γι' αυτό με τα χαρά θα ακούσω την παρουσίαση του κ. Χόισλερ. Όμω από την σκοπιά των συναδέλφων ε, καλό είναι να έχουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, στο δεύτερο ήμιση του πλαισίου, να δούμε πώς τα εργαλεία αυτά μπορούν να προσαρμόζονται για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις του μέλλοντος. Έχω κάποια σχόλια για το θέμα αυτό, αλλά θα προτιμούσα να τα ε, παρουσιάσω μετά την ε, ομιλία του κυρίου Χόσλερ παρά προηγουμένως για να γίνουν καλύτερα αντιληπτά. Ανυπομονώ να ακούσω τον κύριο Χόρσλερ. Ευχαριστώ. Eh bien, nous allons... Euh, Ωραία. Την, την ανυπομονησία σας θα την ευωδώσουμε, ακούγοντας τον κύριο Χόισλερ. Κύριε Διευθυντά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που δίνετε στην Επιτροπή την ευκαιρία να διατρέξει αυτό το τεχνικό ζήτημα, τον προπολογισμό της Γεωργίας και τις σχετικές διαδικασίες. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε την παρουσίασή μας όλα τα βασικά στοιχεία και ζητώ συγγνώμη σε κάποιους από εσά που σας ε, είναι ιδιαίτερα οικεία όλα αυτά τα στοιχεία και μπορεί να σας φανούν περιτά. Προσπάθησα όμως να τα συμπεριλάβω όλα να γίνει μια σφαιρική παρουσίαση για να είμαστε βέβαιοι ότι γίνεται κατανοητό όλο το ιστορικό της διαδικασίας του προπολογισμού. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε απλώς τα δύο βασικά σκέλη της κοινή αγροτικής πολιτικής στον προπολογισμό της. Το Ταμείο το Ευρωπαϊκό Ταμείο των Γεωργικών Εγγύσεων, το EAGF, δηλαδή οι κανονικές πληρωμές και οι δαπάνες της αγοράς. Μιλάμε για μη διαφοροποιημένες πιστώσεις. Κάτι που είναι σημαντικό για τις αιτήσεις συζητήσεις σας περί προπολογισμού. Το δεύτερο στοιχείο είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου. Καλύπτει τα προγράμματα της ανάπτυξης της Υπέθρου και εδώ μιλούμε κυρίως για διαφοροποιημένες πιστώσεις. Κάτι που μοιάζει πολύ με αυτό που ε, υπάρχει ως δομή και στα διευθυντικά ταμεία. Ένα συγκεκριμένο στοιχείο, το οποίο ε, όσο και να το κοιτάξουμε παραμένει το πλέον σημαντικό, είναι τα γενικά στοχευμένα εισοδήματα. Και είναι πολύ σημαντικά για να καθορίσουμε τις αιτήσεις πιστώσεις και τον προπολογισμό. Αυτά τα σηματοδοτημένα, τα στοχευμένα εισοδήματα που είναι ένα εργαλείο του προπολογισμού, ουσιαστικά τροφοδοτούνται από τις ετήσιες διορθώσεις, από παρατυπίες στο παρελθόν. Οι δασμοί του γάλακτος ήταν πολύ σημαντικοί προηγουμένως. Πέρσι, αν θυμάστε, έφταναν τα 8 εκατομμύρια ευρώ και βεβαίως και το πλεόνασμα από προηγούμενους προπολογισμού από προηγούμενα έτη. Αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζουμε τον προπολογισμό. Αυτό που κάνουμε στην έναρξη τη διαδικασίας είναι ότι κοιτάζουμε τις ανάγκες. Κοιτάζουμε τι χρειαζόμαστε για ένα έτος προπολογισμού κατά τη διάρκεια κατάρτισης του σχεδίου και από εκεί αφαιρούμε τα σηματοδοτημένα εισοδήματα για να προχωρήσουμε στη διαδικασία και πολλές φορές είναι σημαντικός ο αντίκτυπος στις πραγματικές ανάγκες. Και λαμβάνονται υπόψη και στις δικές σας συζητήσεις. Για την δημοσιονομική διαχείριση. Μια σύντομη ματιά στο EAGF. Έτσι θα το ονομάζω από εδώ και εξής να σας επισημάνω αυτά τα σημαντικά στοιχεία και την ιδιαιτερότητα του προπολογισμού της ΚΑΠ. Το έτος του προπολογισμού δεν είναι ημερολογιακά καθορισμένα και αυτό απασχολεί και σας όταν ε, εγκρίνετε το σχέδιο προπολογισμού για ένα έτος. Ξέρετε περίπου πώς λειτουργεί το σύστημα. Τα κράτη-μέλη πληρώνουν δικαιούχους βάσει αυτών των πληρωμών κάνουν σχετικές δηλώσεις και η Επιτροπή επιστρέφει τις δαπάνες των κρατών μελών, τις πληρωμές που έκαναν δηλαδή σε συγκεκριμένους μήνες. Επειδή βέβαια όλα αυτά παίρνουν χρόνο, υπάρχει μια διαφορά τριμήνου μεταξύ του πότε πληρώνουν, ε, πληρώνουν τη γεωργοί και πότε παίρνουν πίσω τα χρήματα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως το φθινόπωρο, διότι το φθινόπωρο καταρτίζουμε τη διευθυντική επιστολή τον Σεπτέμβριο και ως τον Σεπτέμβριο δεν έχουμε ακόμη όλες τις τελικές πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες δηλώσεις που πάνε από την 1η Σεπτεμβρίου ως τις 15 Οκτωβρίου. Α, τότε είναι που κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο υπάρχει ένας βαθμός απογοήτευσης και σύγχυσης, διότι δεν μπορούμε στη διευθυντική επιστολή να ε, συμπεριλάβουμε αυτά τα στοιχεία, διότι ε, αυτά τα διαθέτουμε μόνο στις 27 Οκτωβρίου και όχι νωρίτερα. Είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά είναι σημαντική διευκρίνηση, διότι έχει και πολιτικές προεκτάσεις στη διαδικασία συνδιαλλαγής. Διότι ακριβώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ξέρετε ότι έχουμε συστηματικές συζητήσεις μαζί σας, ε, μια φορά το μήνα τουλάχιστον, το λεγόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την εκτέλεση των ποσών μηνιαίως. Τώρα, λίγα λόγια για το Ταμείο της Ανάπτυξης της Υπέθρου. Εδώ το σύστημα είναι κάπως διαφορετικό, διότι έχουμε μόνο τρίμηνιες δηλώσεις, με την ιδιαιτερότητα ότι το τελευταίο τρίμηνο αντικείμενο δήλωση πηγαίνει στον προπολογισμό νη 1. Αυτό έχει προφανώ επιπτώσει και στη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού. Τώρα για το σχέδιο προπολογισμού 2018, μια πολύ σύντομη ενημέρωση. Οι ανάγκε υπολογίζονται σε 11,8 δισεκατομμύρια σε πληρωμές και είμαστε σε ταχύτητα κρουαζιέρας όπως λέγεται. Το πρόγραμμα για τη νέα περίοδο λειτουργεί εύρυθμα και απλώς αυτά τα ποσά είναι περίπου μοιρασμένα κατά 50% σε ετήσια μέτρα, γιατί για την ανάπτυξη της υπαίθρου υπάρχουν μέτρα τα οποία μοιάζουν πολύ με τις άμεσες πληρωμές, για γεωργικά, οικολογικά προγράμματα, για γεωργούς που αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση, ε, για σταθερότητα των τιμών. Αυτά προβλέπουν μια ε, ορατότητα που μας διευκολύνει στη διαδικασία του προπολογισμού. Το άλλο 50% είναι για τα λεγόμενα μέτρα ε, πολιετούς χαρακτήρα. Δηλαδή, παρόμοια δομή με τα διευθυντικά ταμεία. Στην αρχή της περίοδου χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να ξεκινήσουν να αποδίδονται και μετά με τον κανόνα N 3 πάνε κανονικά στο ρυθμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ένα διάγραμμα που φαίνεται φοβερά περίπλοκο, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλούστατο. Θέλω να δείτε απλώ τα χρώματα. Τα χρώματα ορίζουν τις αλλαγές της ΚΑΠ μέσα στις δεκαετίες. Το κίτρινο και το κόκκινο είναι τα παλιά μέτρα της ΚΑΠ, αν μπορώ να τα ονομάσω έτσι, μέτρα της παλιάς ΚΑΠ, εξαγωγικές επιστροφές και παρεμβάσεις στην αγορά. Αρχικά αυτό αφορούσε η ΚΑΠ. Εάν δείτε τώρα τις πρόσφατες εξελίξεις και το σταθερότερο πλαίσιο από το 2007, τα περισσότερα υπερτερεί το πράσινο μάλλον, δηλαδή τις άμεσες πληρωμές, Μερικά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της υπαίθρου και αυτά καλύπτουν το μεγαλύτερο όγκο της ΚΑΠ και των δαπανών της. Αυτό είναι ένα μήνυμα που είναι καλό να επαναλαμβάνεται πάντοτε, διότι δείχνει ότι η πολιτική έχει αλλάξει προ... κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο διάγραμμα αυτό, το οποίο θέλω να το ε, εντοπίσω. Δίνει την εντύπωση ότι αυξήθηκε ο προπολογισμό και θα έπρεπε να υπάρχει εκεί μια διευκρίνηση, αλλά το λέω τώρα προφορικά. Ε, η αρχική κατάσταση ήταν ότι η ΚΑΠ ήταν 70% και παραπάνω του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Στο τέλος της περίοδου αυτής θα έχουμε φτάσει το 34%. Η αύξηση ε, σε αριθμούς ε, σχετικούς αντικατοπτρίζεται από την ε, καταναλογία μείωση της ε, βαρύτητας του προπολογισμού της ΚΑΠ στην όλη κοδόμηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Επόμενη διαφάνεια. Ο κύκλος, το κέικ που δίνει τα μερίδια, της φέτες της ΚΑΠ. Αυτό είναι αντικείμενο διαθεσμικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου μέχρι το 2020 και το μερίδιο συνολικά της ΚΑΠ είναι 38%. Ε, Όπω είπα, 34% προηγουμένω είναι το τέλο τη περίοδου. Υπάρχει μια σταδιακή μείωση, για την ώρα είναι 38% και βλέπετε και τα άλλα σημαντικά κομμάτια του κύκλου στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν έχετε κατά νου αυτούς τους δύο αριθμούς 177 για τα μέτρα της αγοράς και τα υπόλοιπα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, αυτά αλλάζουν ελαφρώς την επόμενη διαφάνεια. Διότι, όπως θα θυμάστε, τα κράτη-μέλη είχαν δυνατότητα να μεταφέρουν από τον ένα πυλώνα στον άλλο αυτό που θα δείτε λοιπόν εδώ σε αυτούς τους ε, λεπτομερέστερους αριθμούς είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων μεταφορών που έχουν ληφθεί από κάτι μέλη. Ίσως χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, απλώς να σας πω για το 2014 βλέπετε πολύ χαμηλό αριθμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου, το EAFRD. Αυτό είναι μια σταθερή τάση που έχουμε και ω διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων προγραμματισμού, θα θυμάστε ότι η απόφαση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ελήφθη μόνο στο Δεκέμβριο του 2013 και το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο άρχισε κατευθείαν την 1η Ιανουαρίου του 2014. Φυσικό το τρόπο λοιπόν υπήρξε αντίκτυπο ε, στην εξέλιξη των προγραμμάτων και ταχύτητα κρουαζιέρας πλοήγησης επετέχθη αμέσω μετά. Να δούμε την ε, υλοποίηση και το που έχουμε φτάσει. Ας πάρουμε μερικές χρονιές στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε πολύ καλή εκτέλεση, ποσοστό εκτέλεση στις άμεσες πληρωμές. Ήδη στον, στην πρώτη χρονιά 97,8%. Πραγματικά είναι πολύ ψηλό ποσοστό, γνωρίζοντας πόσες αλλαγές έπρεπε να καλυφθούν. Περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη ε, βελτίωση το 2018, περιμένουμε ακόμα καλύτερα ποσοστά. Για τις αγορές, σημαντικό να θυμόμαστε τι περάσαμε τα τελευταία χρόνια. Η... Το εμπάργκο στις ρωσικές εισαγωγές, αναταραχές στην αγορά, 1,7 δις προβλέφθηκε για αυτά, καλύπτοντας όλους τους τομείς, κυρίως τα προκυπευτικά, τα γαλακτοκομικά και τα α, ε, κτηνοτροφικά. Απλώς υπενθυμιστικά η κρίση συνδυάστηκε με τη μείωση στα, ε, στις άμεσες πληρωμές ώστε να δημιουργηθεί ένα ταμείο για την αντιμετώπιση της κρίσης εφόσον χρειαστεί που για την ώρα δεν το έχουμε αγγίξει διότι οι πιστώσεις πήγαν αλλού. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για το σκέλος αυτό. Είμαστε αρκετά καλά ως προς το κλείσιμο 2007-2013. 64 προγράμματα περατώθηκαν ως το τέλος του 2016. Και το 2017 έχουμε επιτελέσει ακόμη μεγαλύτερο, μεγαλύτερη πρόοδο. Θα έχουμε κλείσει τα περισσότερα προγράμματα. Ο λόγος που μερικά παραμένουν ανοιχτά, κάποια ζητήματα δηλαδή ανοιχτά, είναι ότι ο κανόνα προβλέπει ότι εφόσον υπάρχει διαδικασία καθάριση για ανοιχτό λογαριασμό σε ένα δεδομένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα δεν μπορεί να κηρυχθεί λήξαν. Άρα Βλέπουμε εδώ πως έχουμε προχωρήσει. Τα περισσότερα από αυτά τα, προβλήματα, τα προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι να λυθεί τελική απόφαση για την εκαθάριση του λογαριασμού. Για τη νέα περίοδο, το 2014 και 2015, έχουμε πάνω από 118 προγράμματα, τα οποία όπως ξέρετε προβλέπουν αιτήσει πληρωμές στους γεωργού για οικολογικά γεωργικά προγράμματα και άλλα και κυρίως επενδύσεις, επενδυτικά προγράμματα που προβλέπεται να κρατήσουν αρκετά χρόνια. Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι αυτό από το οποίο θα μπορούσαμε να ωφεληθούμε από τη στιγμή που οι φορείς πληρωμής, πληρωμών, οι αρχές που έχουν οριστεί στα κάτι μέλη παραμένουν σταθερές στο γεωργικό τομέα. Έχουν διατηρήσει δηλαδή την πιστοποίησή τους και αυτό έχει διευκολύνει εξαιρετικά για να φτάσουμε γρήγορα την ταχύτητα κρουαζιέρας και να προχωρήσουν τα, προγράμματα. Διότι όλοι οι, όλες οι υποδομές στα κάτι μέλη έχουν ε, θεμελιωθεί και έχουν λειτουργήσει σωστά. Ενώ σε άλλα ταμεία που ξέρετε υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Δυσκολίες γιατί κάποιοι από τους φορείς ή τις αρχές δεν λειτουργούν ακόμα ούτε και σήμερα καθώς ομιλούμε. Νομίζουμε λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου προχωρά με καλή ταχύτητα. Έχουμε περίπου 90% των δαπανών ήδη. Μετά το πρώτο τρίμηνο του 2017 είναι υγιές ποσοστό, υγιό, υγιές ποσοστό πρόσληψης των ε, σχετικών ποσών. Τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες για τον πίνακα αυτό, εάν μου επιτρέπετε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να επιστήσω την προσοχή σας στις ανάγκες σε σχέση με τον προπολογισμό το 2017. Θα δείτε ένα μείον, ένα αρνητικό πρόσημο στις δαπάνες για τις γεωργικές αγορές. Μείον 531 ε, ε, ε, εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα γαλακτικών το κομικόν που έχει ανακάμψει και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αίτημα για επιπλέον στήριξη στον τομέα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για την σοβαρή μείωση. τα 247 εκατομμύρια που βλέπετε εδώ ως αλλαγή στις άμεσες πληρωμές για το 2017 είναι ένας ακριβέστερος αριθμός για, τις, για την εκτιμόμενη εκτέλεση στις άμεσες πληρωμές, της εκταμίευσης. το σημαντικό ποσό των 1,7 δις στα, εισοδήμα, στα έσοδα είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων, για, των αποφάσεων εκαθάρισης που περνάνε σε κανονική ταχύτητα. Θα γνωρίζετε ότι είχαμε backlog στις οικονομικές διορθώσεις των κρατών μελών Κάποια δηλαδή πήγαν αναδρομικά και είχαμε κάποια έτη σε πολύ ψηλού αριθμού για μια σειρά ετών. Τώρα επανέρχονται στην κανονική του ταχύτητα. Και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο είχαμε τη σημαντική αυτή μείωση. Επίσης υπάρχει και μια μικρή μείωση στη μεταφορά από τα προηγούμενα έτη προπολογισμού προηγούμενα το 2017. Τώρα, ανακεφαλαιώνοντας περίπου αυτά που είπα, δεν υπάρχει προς στιγμή ανάγκη για περισσότερα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στον τομέα των κτηνοτροφικών. Μικρή που ήδη έχει ψηφιστεί 71 εκατομμύρια για παράταση του τομέα απόσυρσης στα προκυπευτικά μετά τις συνέπειες της ρωσικής κρίσης, στις άμεσες πληρωμές Είμαστε στον ε, συνήθι ρυθμό και ελπίζουμε ο ρυθμός αυτός να παραμείνει σταθερός για το ερχόμενο διάστημα. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν την ευελιξία που τους προσφέρεται για να κάνουν καλύτερη εκτέλεση, έχει και αυτό τις συνέπειες του και θα δείτε μια μικρή μείωση στις ανάγκες, αλλά να έχετε υπόψη ότι δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα, ότι δηλαδή δαπανούμε λιγότερα για αυτό το τομέα, απλώς είναι λιγότερα τα έσοδα που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το 2018 των εσόδων για ειδικό προορισμό βάσει των πληροφοριών που έχουμε προς στιγμή. Για την, ανάπτυξη, για την της υπαίθρου δεν υπάρχουν επιπλέον αιτήματα για το τα 2013 πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις που αναμένονται το 2017 μπορούν να καλυφθούν από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Από το 2014-2020, όπως είπα, είμαστε σε ταχύτητα ρουαζιέρας. Υπάρχει αύξηση του 5,7% που νομίζω ότι μπορούμε να εκτιμούμε ότι θα είναι ο σταθερός αριθμός που θα συναντούμε σε όλο το ερχόμενο διάστημα. Μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά επειδή είναι πολύ πολιτικού χαρακτήρα, υπήρξε συμβολή από το Ταμείο Ανάπτυξη τη Υπαίθρου για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Ένα μικρό ποσό, νομίζω είναι συμβολικού χαρακτήρα, αλλά δείχνει τη σημασία τη πρωτοβουλία ε, αυτή για όλου του χώρου των δαπανών. Αυτό με φέρνει στην τελευταία μου διαφάνεια, η δημοσιονομική πειθαρχία. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η διαδικασία. Θυμηθείτε, 400 εκατομμύρια σε τιμές του 2014 στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο, μέσω της μείωσης των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς, με μια πολύ λεπτομερή διαδικασία που μας λέει μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουμε την πρόταση, μέχρι πότε πρέπει να την έχει δει το Κοινοβούλιο και πότε το Συμβούλιο, καταλήγουμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια διαδικασία light με τη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων. Και φαντάζομαι ότι και εσείς μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Επιτροπή θα λάβει συστάσεις για να την απλουστεύσει. Είναι Μια διαδικασία που ήδη υπάρχει ευρεία συμφωνία, δεν χρειάζεται να είναι ούτε καν τόσο περίπλοκη και μπορούμε να αλλάξουμε και τον αριθμό, διότι ο αριθμός βασίζεται σε πολύ σαφείς υπολογισμούς. Και γνωρίζετε ότι τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται λίγο γιατί είναι ένα εργαλείο δύσκολο να το χειριστούν. Υπάρχουν εξαιρέσεις για τους μικρούς γεωργούς και δεν συμβάλλουν όλα τα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, με λίγα λόγια, αυτή ήταν η επισκόπηση της κατάστασης όπως έχει σήμερα. Ελπίζω να μην ήμουν επιπόλαιος, διότι ε, υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να δώσω περισσότερες λεπτομέρειε και αλλού λιγότερες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή για την παρουσίασή του, η οποία ήταν αρκετά τεχνική Νομίζω ότι αυτό θα καλύψει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, ο οποίος επιθυμούσε να αναβληθεί η ακρόαση αυτή για μετά το καλοκαίρι. Αλλά ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε σαν Επιτροπή και εμείς σαν Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν θέλουμε να εμπλακούμε στην ιεράρχηση των διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων, απλά να μείνουμε σε επίπεδο σεβασμού διαδικασίας. Και έχουμε ανάμεσά μας και εκπροσώπους της Επιτροπής Γεωργίας. Όπως είπατε λοιπόν, κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, δώσατε κάποιες πληροφορίες πολύ χρήσιμες και είπατε ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Θα ξεκινήσω. Λοιπόν, η συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις για όσους το επιθυμούν μέχρι τις 5 και 4 περίπου. Θα ακούσουμε πρώτα 5-6 ερωτήσεις, τις οποίες θα κληθείτε κύριε Διευθυντά να απαντήσετε. Ο πρώτος που θα θέσει η ερώτηση είναι ο κύριος Ashworth. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Χάουσλε. Τρία μικρά σημεία. Πρώτον, κάποια σχόλια. Αν συζητήσαμε για το EAGF και είδαμε ότι έχουν υπάρξει προβλήματα και καθυστερήσεις για τις πληρωμές τους γεωργούς. Θα ήθελα να σχολιάσετε τις καθυστερήσεις αυτές και υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, ανάμεσα στις ε, διάφορες χώρες και ιδιαίτερα σε μία. Δεύτερον, κατάλαβα καλά αυτό που είπατε για τους απλήρωτους λογαριασμούς, που είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και καιρό, ότι η γεωργία και ε, γενικά ο προϋπολογισμός της γεωργίας έχει καλύψει το θέμα αυτό ή όχι ακόμα. Και τέλος, ως εισηγητής για την απλούστευση, η απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής και ως εμπλεκόμενος στην έκθεση των νέων δημοσιονομικών κανονισμών θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας για το θέμα της απλοποίησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και το συγκεκριμένο θέμα είναι η σχέση της γεωργίας και η περιπλοκότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων και των διακανονιστικών ρυθμίσεων. Θα ήθελα να το σχολιάσετε και ίσως ένα τελευταίο σχόλιο. Τον πίνακα. Στον πίνακα βλέπετε πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Ήδη από το 1957 όταν ξεκινήσαμε, τότε ο προϋπολογισμός ήταν το 90% του προϋπολογισμού. Τώρα λέτε και σέβομαι αυτό που λέτε ότι έχει φτάσει στο 34 ενώ νόμιζα στο 38. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για το ποσοστό αυτό του 1% του ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού, των κρατών μελών μάλλον, και συνολικά μιλάμε για 50 περίπου δις. Είναι σημαντικό ε, το θέμα και δεν ξέρω πώς θα επηρεαστεί από το νέο επιπλέον κενό που θα δημιουργηθεί μετά το Brexit, όπου θα έχουμε μια τρύπα γύρω στα 10 δις. Ε, και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, στο μέλλον. Δεν ξέρω αν υπάρξουν ρυθμίσεις τύπου Νορβηγίας ή αντίθετα ε, να υπάρξει επιβολή και από τις δύο πλευρές ε, υψηλού επίπεδου δασμών. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει σημαντικότατο αυτό είναι η κάλυψη των άλλων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα δηλαδή απασχόλησης και ασφάλειας, άμυνας κτλ και εκεί θα πρέπει να υπάρξει αν θέλετε συμπατότητα ανάμεσα στις πολιτικές και τις οικονομικές δυνατότητες. Τρεις είναι οι βασικές λειτουργίες της ΚΑΠ. Καταρχάς, διασφάλιση ε, με ε, αηφόρο τρόπο τροφίμων για 350 εκατομμύρια κατοίκους, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο. Επίσης απαιτείται να υπάρξει και ε, τεχνική πρόοδος στην συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πρέπει να βρούμε τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και ο ισχύων μηχανισμός χρηματοδότησης δεν είναι θα έλεγα συμβατός ε, με τις προκλήσεις. Οι άμεσες πληρωμές μπορεί να φτάνουν και το 20%. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα σε, αυτή, αυτό το ποσοστό και στα άλματα τα οποία απαιτούνται στην παραγωγικότητα. Υπάρχει από την άλλη όμως σχετικά καλή σχέση ανάμεσα στις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν στην γεωργική παραγωγή. Νομίζω λοιπόν ότι και η άμεση στήριξη που είναι ένα μέσο, εν πάση περιπτώσει θα έλεγα άκομψο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να καλυφθούν οι ανησυχίες των επιμέρους μελών που θα θυγούν από τις αλλαγές αυτές. Επίσης ταυτόχρονα οι εγγυήσει ή οι απαιτήσει οι περιβαλλοντικές ποικίλουν και έχουν διαφορετικό ίχνος και επίπτωση από περιοχή σε περιοχή και ιδιαίτερα στον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα έτσι ώστε να επαληθευθεί η επίδοση της κάθε χώρας και δεύτερον να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση και από πλευρά των ίδιων των κρατών μελών, κάτι το οποίο εν μέρη θα καλύψει κάποια από τα κενά. Υπάρχει επίσης το θέμα της διαχείρισης φαινομένων όπως οι ασθένειες και στον φυτικό τομέα και στον ζωικό τομέα και επίσης η αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των τιμών, τα ε, επίσης λεγόμενα υβριδικά μέσα για την αντιμετώπιση των αγορών και για την εξοικονόμηση δαπανών στην κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, ο δείκτης λαθών του ελεγκτικού συνεδρίου είναι αντίστοιχος με την περιπλοκότητα των διακανονιστικών διατάξεων της γεωργίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε. Τώρα δεν περιμένω να μου απαντήσετε σε όλα αυτά, απλά κάνω κάποια σχόλια και θα ήθελα να ακούσω από πλευρά σας ε, να μου πείτε πώς κάποια τέτοια μέσα μπορεί να αλλάξουν έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της ΚΑΠ καλύτερα. Ευχαριστώ τον κύριο Άσουερθ. Αντιμετωπίσατε και τα τεχνικά θέματα και προχωρήσατε επίσης και σε επίπεδο θα έλεγα πολιτικών επιλογών. Είναι πολύ μεγάλα τα θέματα αυτά το θέμα είναι πως μπορεί να καταστήσει κανείς την κοινή αγροτική πολιτική πραγματικά μια σωστή πολιτική, σωστά γεωργική και πραγματικά κοινή. Το 2006 έθεσε σε δοκιμασία σκληρότατη τα έσοδα των γεωργών. Ο κύριος Ντονανό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συνεχίσω αυτά τα οποία έλεγε ο Άσχορθ για την ανταγωνιστικότητα και την απλούστευση των διαδικασιών. Βλέπουμε ότι είμαστε πολύ μακράν της απλοποίησης την οποία θα επιθυμούσαμε. Αυτό δεν αρκεί ούτε για μια τελή πολιτική όπως η δική μας. Ε, υπάρχει το ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν, υπάρχει όμως και το εθνικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει σωστότερος διαχωρισμός του επίπεδου ευθύνης των μεν και των δε και να διασφαλιστεί καλύτερος διάλογος ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα. Και αυτά είναι θέματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Τώρα για τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές σε ορισμένες χώρες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στη Γαλλία είναι τρομερό το πρόβλημα για πάρα πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Υπάρχει μια προσμονή από πλευρά των γεωργών και πολλοί γεωργοί στην ουσία πιστεύουν ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι οι επιδοτήσεις που λένε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι το βλέπουν. Εάν δεν υπάρχει όμως ούτε και αυτό αν δεν έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδά τους μετά τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους, της γεωργικής, τότε κανένας νέος δεν θα εγκαθίσταται πλέον στην γεωργία. Τώρα για τον δεύτερο πυλώνα. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στις διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ περίπλοκες και σε περιφερειακό επίπεδο από ό,τι γνωρίζω όταν λαμβάνει υπόψη κανείς το πώς ε, τέθηκε σε ισχύ ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ με όλους τους ελέγχους εξάντε και εξ ε, δεν τελειώνει ποτέ η διαδικασία αυτή. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία και να επιταχυνθεί η κίνηση. Επί της ουσίας τώρα, και αυτό το είπε και ο κύριος Ashworth θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στον τομέα της ΚΑΠ να επιτρέψουμε στους γεωργούς να ξεπεράσουν και τις υγειονομικές κρίσεις και επίσης τις κλιματολογικές κρίσεις, όπως επίσης και τις διακυμάνσεις ή την πτυτικότητα αν θέλετε των τιμών. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει και τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι ανεπαρκή. Μπορεί κάποια από αυτά να είναι χρήσιμα, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά γιατί το πραγματικό πρόβλημα, η ουσία της υπόθεσης είναι η λειτουργία της ΚΑΠ και η απλούστευση των διαδικασιών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Χόισλερ γιατί ήταν πλουσιότατη η παρέμβαση και πραγματικά υπόθηκε και πολλαπλώς ότι ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την παρουσίαση, παρότι είναι τεχνική, δεν γίνεται κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει να δούμε τώρα και τις ε, βασικές προτάσεις και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, κατάρτιση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου του επόμενου. Και σίγουρα έχουμε και επικοινωνία με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Πρόσφατα δε έγινε και η ανδιάμεση αξιολόγηση του τρέχοντος πολιετούς. Για μένα, εκτός των τεχνικών πτυχών, των αμυγός τεχνικών πτυχών, νομίζω ότι είναι και η σωστή χρονική στιγμή να διαρωτηθούμε τελικά εμείς τι θέλουμε να πετύχουμε και τι μπορούμε να πετύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Αυτό είναι σαφές. Σίγουρα όταν είμαστε βέβαια σε αφηρημένο επίπεδο συμφωνούμε, αλλά συγκεκριμένα πρέπει να πούμε ακριβώς ε, πάνω σε τι θα βασιστούμε. Και νομίζω ότι ε, δεν είναι, είναι μάλλον κοντόφρο να πούμε ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες να το περισσότερες τομείς και περισσότερα κεφάλαια, αλλά ταυτόχρονα λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν λειτουργήσε μέχρι τώρα, δεν θα λειτουργήσει και στο μέλλον. Και αν έχουμε τη δυνατότητα ε, και μιλάμε με το ελεγκτικό συνέδριο, ε, αν εσείς δείτε και συνομιλήσετε με, τους, ε, με τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου στις περιφέρειες σας, θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το γραφειοκρατικό άχθος. Εγώ παραδείγματος μιλώ με, τις, ε, με το Ελληνικό Συνέδριο της Βάδης Βιρτεμβέρης και εκεί μου λένε ότι πραγματικά υπάρχει τεράστιο γραφειοκρατικό άγχος, άγχος και άγχος για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε και να λάβουμε μια απόφαση. Είτε οι διαδικασίες θα απλουστευθούν, οπότε θα γίνουν διαφορετικά τα πράγματα σε κάποιες χώρες, οπότε θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εντό εισαγωγικών, ή αλλιώς θα βούμε, όχι σήμερα, αλλά κάποια στιγμή να το έχουμε υπόψη και για το επόμενο πολιτές κυρίως, να δούμε πού η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει προσθέμενη αξία. Η ερώτηση προς τον κύριο Χόισλερ είναι εσείς τι τομείς βλέπετε σε ό,τι αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις όπου θα μπορούσε κατά τη δική σας εμπειρία ε, να εντοπιστεί η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος γραφειοκρατικός φόρτος. Πού είναι πιο εύκολο να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και πού είναι πιο δύσκολο γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στις ε, χώρες μέλη. Επαναλαμβάνω σε καμία περίπτωση θα πρέπει να επιβαρύνουμε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά πρέπει να δούμε υπάρχουν κάποια σημεία ε, που δεν θα έπρεπε να τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα αναλάβουν ε, οι εθνικές τοπικές αρχές. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποια κράτη που είναι καθαροί εισφορεί και έρχονται αυτά τα χρήματα στι Βρυξέλλε και έπειτα με πολύπλοκε διαδικασίε γυρίζουν πίσω στα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να πούμε εκεί ότι τα αθνικά κράτη θα μπορούσαν να δίνουν αυτή την ενίσχυση αντί να πηγαίνουν έρχονται τα χρήματα ε, μεταξύ εθνικών πρωτεύουσων και Βρυξελών. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τομά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. Το πρώτο ερώτημα είναι αν μπορείτε να μας εξηγήσετε κύριε Χόισλερ αυτή, αυτό το παθηματικό για κρίσεις. που μπορεί να σας φανεί απίστευτο, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί, δεν κινητοποιήθηκε. Παρότι είχαμε την κρίση με τη Ρωσία, με τα κτηνοτροφικά προϊόντα, με το γάλα. Γιατί δεν κινητοποιήθηκε αυτό το παθηματικό ποιοι ήταν οι φραγμοί, ποια ήταν τα εμπόδια και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα εμπόδια στο επόμενο πολιετές. Τι εμπόδια δηλαδή πρέπει να αρθούν για να διευκολυνθεί αυτή, η χρήση αυτού του αποθεματικού για ε, περιπτώσει κρίση. Το δεύτερο, ο Επίτροπος Έτιγκερ μας παρουσίασε το έγγραφο προβληματισμού για το μελλοντικό πολιετέ. πλαίσιο και εκεί υπάρχει κίνδυνο επανακρατικοποίηση τη ΚΑΠ. Μεταξύ των επιλογών αναφέρεται και η επανακρατικοποίηση τη ΚΑΠ. Σε ένα πρώτο χρόνο θα μπορούσε κανείς να πει γιατί όχι. Αλλά σε ένα δεύτερο χρόνο ρωτώ και εσά και ρωτώ με και εγώ. Τι κινδύνους ε, ενέχει μια τέτοια επανακρατικοποίηση. ποιε θα ήταν οι επιπτώσει, ποιε θα ήταν οι συνέπειε στο πλαίσιο μια ενιαία αγοράς όταν οι κρατικές ενισχύσεις ε, θα είναι κρατικές ακριβώς και όχι εθνικές. Συγγνώμη και όχι ευρωπαϊκές. Άρα μπορεί να δημιουργηθεί μία διατάξη της ισορροπίας. Και έχουμε δει αντίστοιχα προβλήματα στο κοινωνικό τομέα ή το φορολογικό. Et juste une petite remarque, mais qui ne concerne pas και ένα τελευταίο σχόλιο που δεν αφορά την Κομισιόν, αλλά εμά. Καταλαβαίνω τους συναδέλφου που θέλουν πιο μεγάλη απλούστευση. Όταν όμως η Κομισιόν προτείνει μια έκθεση omnibus για την απλούστευση, ορισμένοι από τους συναδέλφου ε, δεν διστάζουν να καταθέσουν τροπολογίε ώστε τελικά να μην έχουμε τόση απλούστευση. Ευχαριστώ την κυρία Τομάλη, ο Πρόεδρος που μας επισήμανε και τις αντιφάσεις μας. Φυσικά και ως καινούργιο ζητάμε συνεχώς ε, την απλούστευση, αλλά ταυτόχρονα λόγω τελειομανίας με τις ε, ε, τροπολογίες μας δεν πάβουμε να κάνουμε ακόμα πιο πολύπλοκους κανόνες από την άλλη πλευρά. Πώς θα τα εφαρμόσει όλα αυτά η Κομισιόν μετά που τη ζητούμε. <laughs> La parole est à Madame la Présidente le Κύριε Πρόεδρο Γκρέσλιχ τώρα το λόγο συνεισηγητρία με τον κύριο Άσουερθ για τα θέματα απλούστευσης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, αλλά είχα δύο ομάδες επισκεπτών και δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν. Όλοι παραπονόμαστε για τους ε, ελέγχους και ιδίω για τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Το έχουμε και στην Επιτροπή μας το όνομα αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι τόσο το πρόβλημα δεν είναι ο έλεγχος του προϋπολογισμού, ο δημοσιονομικός έλεγχος, αλλά η τεχνική έλεγχη και η ουσιαστική έλεγχη στον τομέα της γεωργίας είναι το θέμα. Έχουμε 16 κανονισμούς, ε, την πολλαπλή συμμόρφωση και τους, κανονισ... τους έλεγχους μάλλον που θέλουν να, να αποδείξουν ότι παρμόζονται βέλτιστες πρακτικές. Έχετε μπει στον κόπο εσείς ε, ως Κομισιόν να δείτε πόσους δημοσιονομικούς ελέγχους έχουμε στον τομέα της Γεωργίας και πόσους ε, ουσιαστικούς τεχνικούς ελέγχους. Καλώς. Ο πρόεδρος δεν βλέπω κάποιον άλλον θέλει το λόγο. Θα παρακαλέσω λοιπόν ε, να μας απαντήσει ο κύριος Χάσλα, αφού εγώ πρώτα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όταν ε, προετοιμάζουμε το επταετές πολιετές μας πλαίσιο, πώς προχωράμε, πώς κάνουμε την ε, κατανομή των κονδυλίων ανακράτος μέλος. Γιατί πέραν των άμεσων ενισχύσεων, οτικοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τι ε, δικαιούται το κάθε κράτος και κάθε κράτος έπειτα φροντίζει να επαληθεύσει κατά πόσον έλαβε το μερίδιο που προβλεπόταν να λάβει. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ακριβώς πώς έχει η διαδικασία ε, προετοιμασίας του πολιετούς δημοσιομικού και της ε, κατανομής των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω ένα παράδοξο γιατί ουσιαστικά ε, στηρίζουμε τα γεωργικά εισοδήματα, όμως αυτά προκύπτουν από τις τιμές. Και οι αγρότες θα ήθελαν να υπάρχει μια ισορροπία. Όχι με επιδοτήσεις, αλλά με τιμές. Και λόγω των ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, πολλέ φορέ μειώνονται οι τιμέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνίε που συνάπτουμε εμεί. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιε οικονομίε ε, με την κοινωνική πολιτική, ακολουθώντα ένα διαφορετικό όραμα σε ό,τι αφορά τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά δε και το κομμάτι που αφορά τα γεωργικά προϊόντα σε αυτέ τι συμφωνίε. Επίσης, η Ευρώπη παγορεύει κανονισμούς, βάζει απαγορεύσεις παρακολουθάει στα ζυζανιοκτώνα. Όμως, αν απαγορεύουμε κάποια προϊόντα, η γλυφοζάτη για παράδειγμα, τα νεονικοτινοειδή κτλ δεν θα έχει η ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Ένωση το καθήκον να χρηματοδοτεί την έρευνα για να προτείνει εναλλακτικά προϊόντα τα οποία δεν θα υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Αυτές είναι οι δικές μου ερωτήσεις. Οπότε, τώρα ο λόγος σε εσά, κύριε Διευθυντά, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με βάζετε σε δύσκολη θέση. Γιατί εγώ ήρθα εδώ έχοντας υπόψη ότι θα έχουμε μια τεχνική ανταλλαγή απόψεων για τα δύσκολα ζητήματα που άπτονται του προπολογισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ακούστε, ε, τα ακούω και στην εκλογική μου περιφέρεια και φαντάζομαι και οι συναδελφοί μου το ίδιο. Είναι τόσο πολύπλοκο γιατί μιλάτε για τεχνικά θέματα που άντε να εξηγήσει ε, στου δικαιούχου πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Και όταν είναι τόσο πολύπλοκη μια πολιτική που δεν μπορεί να την εξηγήσει, πάβει να είναι και πολιτική. Άρα, χάρη και στην κυρία Γκρέσλε, θα πρέπει να βρούμε τα στοιχεία αυτά που θα οδηγήσουν σε απλούστευση, αλλά πραγματική απλούστευση. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το μόνο μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι ουσιαστικά ο κύριος Χόγκαν ή ένα ε, γενικό διευθυντή. Ε, ο γενικός διευθυντή γεωργία θα πρέπει να είναι εδώ για να σα απαντήσει στα τόσο πολιτικά αυτά ζητήματα. Ε, ΕΕ. Παρ' όλα αυτά, να προσπαθήσω να σχολιάσω. Με τον κύριο Άσχορεφ πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι Ουσιαστικά αναφέρατε στην παρέμβασή σας όλα τα πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα που μας απασχολούν και που είναι υποσυζήτηση. Και όπως γνωρίζετε, ο Επίτροπος Χόγκαν έχει υποσχεθεί για αργότερα φέτος ε, μια ανακοίνωση για τον εξυγχρονισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν τα οποία εσείς θέσατε θα είναι αντικείμενο αυτής της ε, διαδικασίας. Για να μπω σε λεπτομέρειες. Μιλήσατε για τις ε, προθεσμίες ε, και κυρία Τωμά νομίζω, για τις προθεσμίες πληρωμών. Όχι, δεν ανώ. Αυτές οι προθεσμίες, αυτές οι διορίες για τις πληρωμές ε, είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά και όχι και τόσο τεχνικό από την άλλη πλευρά, γιατί αν θυμάμαι καλά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό που πάντοτε επέμενε να υπάρχουν προθεσμίες στην νομοθεσία σε σχέση με τις πληρωμές. Όταν θα πρέπει δηλαδή να δίνονται κάποια χρήματα στους αγρότες. Και αν θυμάστε καλά, ε, στο προηγούμενο πολιετές ήταν πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου να μπουν και για το δεύτερο πυλώνα προθεσμίες για τις πληρωμές. Δεν είναι δηλαδή τα κρατημέλη αυτά που θα αποφασίζουν πότε θα μπορούν να πληρώσουν τους αγρότες. Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, συγκεκριμένες διορίες ε, και αν δεν τις εκπληρώσουν, αν δεν τις στηρίσουν, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη. Και το κράτος μέλος που γνωρίζετε καλύτερα από τα άλλα, κατά το παρελθόν, έγινε αντικείμενο σοβαρών διορθώσεων, σοβαρών δημοσιονομικών Διορθώσουν που έπρεπε να τι αποδεχθούν επειδή δεν είχαν πληρώσει εγκαίρω του αγρότε. Υπάρχουν λόγοι για του οποίου πρέπει να δεχθούμε και το ξέρετε για πέρυσι και ε, αφορά και τη Γαλλία. Υπήρχαν και άλλα κρατημέλη όμω που ήταν στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή καθυστέρησαν τι πληρωμέ για του ε, γεωργού επειδή ήταν η πρώτη χρονιά τη ε, μεταρρύθμιση, τη νέα μεταρρύθμιση. Υπήρχαν λοιπόν ζητήματα και με τα συστήματα πληροφορική αλλά και με άλλα συστήματα και μισοσκομισιών δείξαμε κατανόηση φυσικά, γιατί δεν είχαμε κανένα συμφέρον να βιαστούν, να πληρώσουν ε, τα κράτη-μέλη, αλλά με πάρα πολλά λάθη και τελικά να υπάρξει πλήρη σύγχυση και χάος. Γι' αυτό και παρατείναμε αυτές τις ε, διορίες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα θέματα και είναι κάποια από αυτά εκτός ελέγχου των κρατών μέλων. Αν ένα κράτος μέλος όμως έρθει πολύ απλά και μας πει τώρα την 11η ώρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το σύστημα πληροφορικής, ε, αυτό δεν είναι και λόγος για να τους επιτρέψουμε να πληρώσουν με καθυστέρηση τους αγρότες. Το θέμα είναι οι αγρότες να παίρνουν εγκαίρω τα χρήματα. Αυτό είναι το θέμα. Όχι να βοηθούμε τις διοικήσεις να λύσουν τα προβλήματά τους. Επίσης, σύντομα ασχοληθήκατε με τα ράλ, τα υπόλοιπα προς ακαθάριση ανεξόφλητο λογαριασμό στο δεύτερο πυλώνα. Δεν είναι πρόβλημα και το επιβεβαιώνω. Στο δεύτερο πυλώνα πάρα πολύ μικροί ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Πάμε πολύ καλά με το κλείσιμο, άρα δεν, υπάρχουμε, δεν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι σε ό,τι αφορά δηλαδή, την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Απλούστευση είναι ένα άλλο θέμα. Όλοι νομίζω το αναφέρατε όσοι πήρατε το λόγο. Πράγματι, κάναμε μια πρόταση πρόσφατα και όπως ξέρετε εγκρίθηκε και μια κατεξουσιοδότηση πράξη για τη μεταρρύθμιση, την οποία ψηφίστηκε πριν από κάποιε εβδομάδες στο Κοινοβουλίο και περιλαμβάνει σημαντικά ε, μέτρα απλούστευση. Έχουμε και την πρόταση Omnibus που είναι υποσυζήτηση και για τη Γεωργία επίσης ένα πυλώνας είναι η απλούστευση και ελπίζω να έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Όμως, το γενικό ζήτημα που όλους σας απασχόλησε νομίζω ασκεί όλο και περισσότερη πίεση στην ε, πολιτική γεωργία. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα, ο κύριος Χόγκαν, ο Επίτροπος, ε, το έθεσε ως προτεραιότητα. Ότι δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια ουσιώδη ζητήματα στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής, ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το φαύλο αυτό κύκλο. Να υπάρξει μια νέα διάταξη. Να έχουμε νέα κριτήρια επιλεξιμότητας Κύριο Σαρτούη διακόπτη. Θα ήθελε κυρία Γκρέσλε να κάνει μια παρατήρηση ίσως και να σας ε, διατυπώσει ένα ερώτημα. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα στο Στρασβούργο, συμμετείχα στι διαπραγματεύσει Επιτροπή Γεωργία, στον τριμερή διάλογο δηλαδή, σε ό,τι αφορά το Omnibus και το τμήμα που αφορά τη Γεωργία. Και υπήρχαν και κάποιε τροπολογίε Επιτάπητο. σε σχέση με τα εκτάρια. Για το Land Identification System έχει δεκασαπλασιαστεί το, το συγκεκριμένο νούμερο. Είναι 10 εκτάρια τώρα. Τα κράτη που είχαν ένα σύστημα που λειτουργούσε τιμωρούνται και επενούνται ή τέλο πάντων επιβραβεύονται αυτά που δεν είχαν. Άρα, ο δεκαπλασιασμός αυτής της επιφάνειας ε, από ε, σχεδόν ένα εκτάριο να είναι δέκα, ε, πού οδηγεί σε απλούστευση. Αυτή είναι η ερώτηση. Για το συγκεκριμένο αυτό σημείο. Ήταν 0,1 και έγινε 10. Στα περισσότερα κράτη-μέλη διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια μονάδα μέτρησης που να επιτρέπει, κάποιο μέγεθος που να επιτρέπει μηδενικά περιθώρια σφάλματος. Αυτό ήταν το θέμα. Ο στόχος είναι να μην παίρνουν οι αγρότες ε, πολύ μεγάλες ενισχύσεις για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Αλλά νομίζω ότι παραμένει σε ένα επίπεδο ε, λογικό αλλά εσείς εδώ έχετε αναφέρει ένα πολύ λεπτό ζήτημα, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλά κράτη που ε, είναι ότι δεν υπήρχαν μεγάλα προβλήματα για πολλά κράτη-μέλη με την εφαρμογή της ε, νέας αυτής διάταξης και το ελεγκτικό συνέδριο φέτος σε ένα πολύ μεγάλο τομέα, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις, ε, νομίζω ότι θα δώσει δήλωση αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή αυτές οι προϋποθέσεις και αυτό η τάξη μεγέθους έχουν τεθεί και πρέπει να εφαρμόζονται. Το θέμα είναι όμως ποια είναι η τιμή. Για να επιτευχθεί αυτό ο αυτή η προϋπόθεση. Δικαιολογείται, αιτιολογείται και αν μου επιτρέπετε, επειδή και εσείς κάνατε μια ερώτηση, που είναι τα περισσότερα που έχουμε τις περισσότερες τέτοιες υποθέσεις στον πρώτο και στον δεύτερο πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα τα κράτη-μέλη έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες, ενώ στον πρώτο ορίζονται πολύ περισσότερα από τις Βρυξέλλες. Άρα τα λάθη γίνονται στον πρώτο. Στο δεύτερο πυλόν έχουν πολύ μεγάλο περιθώρια τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές για να εφαρμόσουν ε, τα μέτρα που θέλουν. Βέβαια θα πρέπει να βλέπουμε και το θέμα του κόστους και το θέμα της αναγκαιότητας αυτών των μέτρων. Υπάρχει και το λεγόμενο gold plating, όπως λέμε εμείς εδώ στις Βρυξέλλες, αυτός ο υπερθεματισμός, ε, ο κανονιστικός που πολύ συχνά οδηγεί να νιώ, τον γεωργό, τον κοτρινοτρόφο ή τον δικαιούχο να νιώθει ότι ελέγχεται, ότι τον παρακολουθούν και τον ελέγχουν συνεχώς ε, οι ελεγκτικές αρχές ε, και από τις Βρυξέλλες. Και σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση, αυτό είναι και από τα σημαντικά ερωτήματα και προβλήματα, το ουσιαστικό δίκαιο δηλαδή, που δεν έχει να κάνει με τη γεωργική πολιτική και τη γεωργική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τους κανόνες που ισχύουν για τις ε, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για τους αγρότες, ε, που ισχύουν για τους δικαιούχους των ενισχύσεων. Και εντάξει, υπάρχει ανάγκη για αυτούς τους ε, κανόνες και προϋποθέσεις, όμως πραγματικά όλα αυτά ενισχύουν την εντύπωση ότι ο δικαιούχος είναι περικυκλωμένος από ελεκτικές αρχές και δεν μπορεί πλέον να κάνει τη δουλειά του. Αν με επιτρέπετε τώρα να πω τα υπόλοιπα στα αγγλικά, γιατί δεν απάντησα εντελώς τον κύριο Άσχουερθ. Δέχεστε να σας διακόψει ο κύριος Κέλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα κύριε Χόσλε γιατί σας έδωσε ένα παράδειγμα η κυρία Γκρέσλερ από την ε, ανοχή αυτό το ποσοστό που δεκαπλασιάζεται ε, από που προκύπτει αυτή η απλώστευση. Ποια είναι η οριακή τιμή, για πόσα χρήματα μιλάμε, για τον, είναι, αν ήταν 300, συγγνώμη, αν ήταν ένα ε, εκτάριο 300 ευρώ. Δηλαδή από 30 πάμε στα 300 ευρώ. 12 εκατομμύρια ετησίως παραπάνω για την ΚΑΠ. Ναι γιατί στρογγυλοποιούμε ανεκτάρι. Το πρόβλημα που έγκυται. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκπίπτουν ε, του υπολογισμού όταν είναι κάτω από το ένα εκτάριο. Αυτοί που είναι πάνω από το εκτάριο μπαίνουν στην ίδια κατηγορία. Άρα δεν έχουμε μείωση του διοικητικού άκθους, αλλά το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Το θέμα είναι να έχουμε επιλέξει μια τάξη μεγέθους ώστε να μπορούν οι αγρότες να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι το σημαντικό και όχι ακριβώς ε, πόσο είναι το εκτάρια. Wird jetzt gar nicht erwartet, dass ich so schnell dran komme. Also. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, ο κ. Γκάιερ. Και επανέλθω σε αυτό που είπε ο κ. Σκέλμελ. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός κίνδυνος. Μέχρι 300 ευρώ γεωργική εκμετάλλευση. Το είπε και η κυρία Γκρέσλε. τελικά έχουμε μείωση του διοικητικού φόρτου ή όχι. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί εγώ νομίζω πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να τα ξεκαθαρίσουμε. Τα δύο δεν μπορούμε να τα έχουμε, ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, είτε δεχόμαστε μια κάποια βεβαιότητα σε ό,τι αφορά το ύψος του ποσού που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν ήταν και τόσο καλή η ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρότι ήταν καλοπροαίρετη σε ό,τι αφορά το ανεκτό ποσοστό σφάλματος που είναι σαν να λέμε «Ε, δεν μας πολύ νοιάζει και κοιτάμε από την άλλη πλευρά αλλά τελικά η βασική δεν είναι σωστή. πόσους έλεγχους θα κάνουμε για να βρούμε ε, σφάλματα τα οποία κινούνται σε μια περιοχή που δεν δημιουργεί ε, ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή να δαπανίσουμε 10.000 ευρώ για να βρούμε ένα σφάλμα τη τάξη των 10 100 ευρώ. Αυτό εννοώ. Οικονομικά δηλαδή δεν έχει ε, νόημα κάτι τέτοιο. Και πώς θα το εξηγήσουμε στους Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Αν ε, το κάνουμε αυτό, θα έχουμε τα ελεγκτικά συνέδρια σε διοικητικό επίπεδο που θα πρέπει να τα επαληθεύσουν όλα, σε τοπικό επίπεδο. Τελικά ο αγρότης επιβαρύνεται ή όχι. Γιατί είναι η επιλογή, ελέγχουμε τα πάντα, οπότε επιβαρύνεται ο αγρότης ή όχι. Γιατί μπορούμε να φτάσουμε και να ψάχνουμε και το ευρώ και το σέντ το σφάλματος. Οπότε να είμαστε πάρα πολύ γραφειοκρατικοί και να επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες. Αυτό το λάβουμε υπόψη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το συζητήσουμε και εμείς εδώ. Τι είμαστε έτοιμοι δηλαδή να δεχθούμε. Πόσο, ε, πόσους ελέγχους και με ποιο κόστος ε, θα ε, επιβάλλουμε ή θα επιτρέψουμε τελικά. Γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα, τα σφάλματα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε παρά σε μια ιονή ακρίβεια. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα μας ε, ε, απασχολήσει πάντοτε. Παραδείγματο χάρη υπάρχει ένα ε, χωράφι που μπορεί να έχει όμως 10 δέντρα. Θα πούμε ότι είναι δάσος ή θα πούμε ότι είναι χωράφι. Πάντα θα έχουμε ε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε σκιαμαχία εδώ και να κυνηγάμε φαντάσματα έλεγχοι χρειάζονται και ποιοι είναι αυτοί οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν ε, τη σημασία τους για να εξασφαλίσουν ε, την ακρίβεια. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή στον κέντρινο τύπο θα βγούνε διάφορα άρθρα και μετά θα βγούμε όλοι να αντιδράμε. Ενώ πρέπει να τα δούμε τα πράγματα πιο λογικά. Κύριε Διευθυντά, να απαντήσω στις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Γκέγερ ή να ε, συνεχίσουμε τις ερωτήσεις που είχα σημειώσει από πριν. Να πούμε ότι ο κύριος Γκέγερ ήταν ουσιαστικά η συνέχιση της παρέμβασης της κυρίας Γκρέσλε. Επί της ουσίας, ποια είναι τα μικρότερα ποσά που εκταμιεύονται ε, με την ΚΑΠ αναγεωργό. Υπάρχουν ελάχιστα ποσά δικαιούχοι που παίρνουν κάτι εκατοντάδε ευρώ. Όχι παραπάνω. Ιδίω ορισμένε χώρες με πολύ μικρές δομές. Κάποιοι γεωργοί παίρνουν ελάχιστα ποσά. Ξέρετε ότι η Επιτροπή έχει κάνει προτάσεις για να περιορίσει, να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο για τους δικαιούχους και αυτό διαρκώς το απορρίπτει το Συμβούλιο για λόγους κατανοητούς. Ορισμένες χώρες η κατηγορία των δικαιούχων που παίρνουν ελάχιστα ποσά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. στο σύστημα ε, υπάρχει και μια δυνατότητα πλουστευμένου μηχανισμού κατά αποκοπήν ποσών για να πληρώνονται οι γεωργοί. Υπάρχει, χρησιμοποιείται σε κάποια κάτι μέλη, αλλά ίσως δεν αξιοποιείται παρκώς από όλους όσοι θα μπορούσαν να υποφελούνται. Να ξεκαθαρίσω το εξή. Το σύστημα μας είναι έτσι που για να δώσω το παράδειγμα μας 300 ευρώ. Τι θα πει αυτό το όριο των 300 ευρώ ένα εκτάρι. Κίνδυνος για το ταμείο είναι για το δικαιούχο είναι το 100% της βοήθειάς του αν τη χάσει για το ταμείο μου 300 ευρώ. Εάν ο δικαιούχο ξεπεράσει τα χ εκτάρια που έχουμε λάβει ως ε, σημείο αναφοράς για το σεβασμό του κανονισμού, εάν το ξεπεράσει ως ε, γεωργό, είναι σαν την ε, γκυλοτίνα, χάνει σαν τη λεμιτόμο. Χάνει όλο το ποσό. Αυτό δημιουργεί τις δυσκολίε. τα παραδείγματα που μόλι έδωσε ο κ. Γκάγερ. Στην Αυστρία ιδιαίτερος, πριν από τρία χρόνια, Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις ε, βοσκοτόπων ή ε, δασικών εκτάσεων, ε, εκτάσεων με δέντρα, όπου η δασικων εκτασεων εκτασεων με δεντρα οπου η δικη της Επιτροπής, κάνοντας τη μέτρηση, έλαβαν την απόφαση ότι το σύνολο των ποσών που εκταμεύονταν για τους γιοργούς ε, ήταν για περιπτώσεις μη επιλέξιμες. Έτσι είναι το σύστημά μας δεν είναι αν έχεις τόση γη παίρνει τόσο ποσό, όχι. Αν δεν ε, συμμορφούσε με τους κανόνες όπως είναι ορισμένοι, έχουν οριστεί, χάνεις όλη τη βοήθεια. Οπότε χρηματοδοτείται με ο κίνδυνο, σε κάποιε περιπτώσει είναι μεγαλύτερο, αλλά περισσότερο από εκατοντάδε ευρώ για κάποιου. Ε, διότι εάν ο κύριο Στάδε έχει ξεπεράσει την επιφάνεια που του αναλογεί, την έκταση που του αναλογεί, χάνει όλη τη βοήθεια που παίρνει. 500 ευρώ, όσα και αν είναι αυτά. Εκείνη η περιπλοκότητα της πολιτικής φύσης του όλου θέματος. Και καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε κι εσείς ε, να πάρετε την απόφαση, αλλά τα κοιτάζουμε ανά εκτάρια από πολύ κοντά, με το μικροσκόπιο. Συνεχίστε. Να συνεχίσω για να μην ξεχάσω τη σειρά, να πάρω ένα-ένα από τον κατάλογο που τα έχω σημειώσει. Ο κύριος Άσφορθ, για να ξανάρθω σε εσάς. Αναφερθήκατε στο Brexit και κατανοείτε ότι δεν είμαι σε θέση να σας δώσω οποιαδήποτε ένδειξη για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Γνωρίζετε πάντως ότι έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, τα δημοσιονομικά θέματα θα παίξουν σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είμαι φυσικά σε θέσεις και δεν έχω και τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν. Μιλήσατε για τη διαχείριση κινδύνου, το risk management, και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο στα πλαίσια της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής θα βρείτε κάποιες ε, πιο ε, ισχυρές, θα έλεγα, διατάξεις αυτός είναι πράγματι ένας τομέας όπου οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν πλέον διατυπωθεί στο έγγραφο και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ε, για να τις εφαρμόσουμε και να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Ε, να στοχεύσουμε σε μια καλύτερη δυνατότητα βοήθειας προς τους γεωργούς. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε όπως το είχαν προτείνει και προετοιμάσει εν μέρη η κυρία Έτιγκερ και η κυρία Κρέτσου. Είναι κάτι που άρτητε του μέλλοντος της ΚΑΠ, για να έρθω τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Ντενανό. Θα επαναλάβω ουσιαστικά κάτι το οποίο είπα θα υπάρξουν προθεσμίες για τις πληρωμές και για το δεύτερο πυλώνα. Αυτό αποφασίστηκε άλλωστε και στα πλαίσια του δεύτερου πολιετούς δημοσιονομικού, έτσι ώστε να μην περιμένουν πάρα πολλοί γεωργοί. Για την απλοποίηση νομίζω ότι καλύπτεστε από αυτά που είπα προηγουμένως για την πρόταση Omnibus. Ελπίζω να έχουμε βελτιώσει στο ταχύτερο δυνατόν για τον κύριο Κέλμελ σας είπα ότι ο δεύτερος πυλώνας τίνει να υφίσταται βαρύτερους ελέγχους από τον πρώτο πυλώνα. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει στα κράτη-μέλη και στα λέντερ τα γερμανικά. Υπάρχει η αίσθηση ότι τα προγράμματά μας είναι περίπλοκα, επακριβή και απαιτητικά. Πολλαπλά απαιτητικά. Ένα γενικό σχόλιο εδώ. Υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στην περιπλοκότητα και τους στόχους τους οποίους θέτει κανείς. Με άλλα λόγια, υπάρχει αρκετά χαμηλή περιπλοκότητα στις άμεσες πληρωμές, αν δεν μιλήσουμε για το greening, γιατί οι προϋποθέσεις για πρόσβαση στις άμεσες ε, πληρωμές είναι το να έχει κανείς ε, μια κάποια έκταση και αν έχει την έκταση βασίζεται ο υπολογισμός σε αυτό και παίρνει τα χρήματά του. Εν πάση περιπτώσει και με τους δορυφορικούς, τα δορυφορικά μέσα ελέγχεται. Αλλά όσο περισσότερο ζητάει κανείς από έναν δικαιούχο ας πούμε ότι πρέπει να επενδύσει, ότι πρέπει να δηλώνει προμήθειες, ότι πρέπει να καταθέτει επιχειρηματικά σχέδια, πρέπει να κάνει επενδύσεις φιλικές για το περιβάλλον, επενδύσεις που να ανταποκρίνονται στα επίπεδα φυτογίνης που απαιτούνται. Όσο πιο απαιτητικός είσαι, τόσο πιο αντικειμενική είναι η στόχη που θέτεις τόσο καλύτερα στοχευμένη είναι η προσπάθεια που γίνεται, αλλά ο δικαιούχος είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες για να τα πετύχει. Αυτό είναι ένα από τα παράδοξα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Σαν πολιτική θα πρέπει να γνωρίζουμε το τι θέλουμε. Θέλουμε συγκεκριμένους στόχους ή θέλουμε ε, κάποιους απλούς εφαρμόσιμους βέβαια κανόνες. Νομίζω ότι κάθε συζήτηση για την απλοποίηση αυτό θα πρέπει να έχει σαν στόχο. Για την κυρία Τομά, είπατε... Κοιτάξτε, δεν χρησιμοποιήθηκε το αποθεματικό κρίσης γιατί είναι η τελευταία προσφυγή. Αν δεν έχουμε καθόλου χρήματα, στο χρηματοκιβώτιο, τότε μόνο θα τη χρησιμοποιήσουμε. Ευτυχώς ή δυστυχώς παρόλες τις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια πάντα υπήρχαν κάποια χρήματα διαθέσιμα. Και ακριβώς και με τις, τα προδιαγεγραμμένα έσοδα α, οι, υπήρξαν ορισμένες διορθώσεις δημοσιονομικές που έγιναν, υπήρξαν επίσης και κάποιες εισφορές οι οποίες ήταν ανέπαφες, ε, και έτσι πάντα στο κεφάλαιο 2 υπήρχαν κάποια χρήματα διαθέσιμα που μας επέτρεψαν να χρηματοδοτήσουμε τις κρίσεις αυτές χωρίς να προσφύγουμε στο αποθεματικό για την κρίση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα συζητήσετε στα πλαίσια του επόμενου ε, πολιετούς δημοσιονομικού. Τώρα για τους κινδύνους επανεθνικοποίησης τους οποίους αναφερθήκατε. Και εδώ αναφέρομαι στο έγγραφο το οποίο κατέθεσε ο Επίτροπος Έτιγκερ και η Επίτροπος Κρέτσου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρότασή της, δεν πήρε μια τελική θέση και αυτό το οποίο είπατε δείχνει ότι έχουμε ένα σημαντικό επιχείρημα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ποιος είναι ο κίνδυνος πραγματικά της επανεθνικοποιήσεως ε, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας ορισμένα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα και την επιθυμία να συγχρηματοδοτήσουν ενώ άλλες χώρες δεν έχουν ή το ένα ή το άλλο ή και τίποτα από τα δύο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προηγηθούν τη συζήτηση της συγχρηματοδότησης. Εδώ υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού γιατί δεν θα πρέπει να τιμωρούνται οι παραγωγοί στα πλαίσια μιας ενιαίας αγοράς, σαν παράδειγμα, μέσω τέτοιων μέσων τρόπων στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η κυρία Τομά, ε, κοιτάξτε, η ερώτησή μου ακριβώς ήταν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια μελέτη επιπτώσεων, μια μελέτη συνεπειών για την πιθανότητα της μερικής ή συνολικής επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος. Το θέμα της νομιμότητας, του σεβασμού των κανόνων και σε εθνικό επίπεδο είναι οι κανόνες αυτοί ικανοί να αποτρέψουν την εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων. Μία από τις δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσετε είναι ότι μπορεί να προβλέψετε κάποιους κανόνες εθνικών επιδοτήσεων που δεν επιτρέπουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Μπορεί να έχουμε όμως κάποιες ρυθμίσεις εθνικές οι οποίες να υποχρεώνουν την χώρα να συγχρηματοδοτεί. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία έθεσαν ακριβώς πρώτων ευθυνών όλων οι δύο επίτροποι στους οποίους προαναφέρθηκα. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, για τις δύο δικές σας ερωτήσεις. Η κλίδα κατανομής. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων του πολιετούς δημοσιονομικού. Πράγματι η συζήτηση γύρω από τη δίκαιη επιστροφή είναι μια από τις ιδρυτικές αν θέλετε αρχές της ΚΑΠ. Υπάρχουν επιστώσεις πολύ συγκεκριμένες οι οποίες διανέμονται για το τμήμα των άμεσων πληρωμών στον πρώτο πυλώνα. Συνεπώς κάθε κράτος μέλος γνωρίζει το δικαίωμα αν θέλετε ίσπραξης εκ των προτέρων 100%. Αυτό δεν εφαρμόζεται στο κομμάτι της αγοράς, το οποίο και αυτό ανήκει βέβαια στον πρώτο πυλώνα, αλλά δεν υπάρχουν ε, διαγεγραμμένα ποσά. Εκεί τα χρήματα εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι τμήμα ε, της πολιτικής συμφωνίας την οποία είχατε προβεί εσείς οι ίδιοι στο Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο για την κατανομή των πιστώσεων. Επιβεβαιώνω λοιπόν ότι για τα κρατημέλη τα πράγματα πρέπει να γίνουν πιο ξεκάθαρα ε, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να έχουν από την κοινή αγροτική πολιτική, κάτι το οποίο είναι σημαντικός παράγων σταθεροποίησης. Κοιτάξτε, ε, μήπως έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό πρόβλημα της δημοσιονομικής πραγματικότητας να δίνουμε χρήματα στους γεωργούς κάτω από συνθήκες κατά τις οποίες δεν έχουν την ανάγκη. Ενώ όταν υπάρχει σοβαρή κρίση, λόγω του ετήσιου χαρακτήρα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων και κάθε χώρα εξαντλεί το σύνολο των πιστώσεων στις οποίες έχει δικαίωμα, καταλήγουμε σε παράλογες καταστάσεις. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τον ετήσιο χαρακτήρα, τον ενιαύσιο σε εισαγωγικά χαρακτήρα, μιας πολιτικής σαν την ΚΑΠ. Είναι δυνατόν να ξεφύγουμε από το χαρακτηριστικό αυτό και να ακολουθήσουμε με πιο εύθετο τρόπο την συγκυρία. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε απόλυτα τεχνικό επίπεδο, αλλά κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Έχετε ένα σύστημα σαν των Ηνωμένων Πολιτειών, σαν παράδειγμα, το οποίο είναι συγκυριακό θα έλεγα. Δεν υπάρχει ένα δικαίωμα ίσπραξης ενώ εμείς καθορίζουμε μονομένα δικαιώματα για κάθε χώρα και για κάθε γεωργό. Κάποιος ο οποίος εκπληρεί τις προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να εισπράττει την επιδότηση αυτή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολιτική υποχρέωση μόνο, είναι δικαίωμα. Αλλά ένα δικαίωμα δεν συνιστά μια πολιτική, λέει ο πρόεδρος Ατουή. Η πολιτική είναι μια σειρά μέσων για να λυθεί ένα πρόβλημα, ενώ ένα δικαίωμα είναι μια αυτόματη πληρωμή. Και γι' αυτό ακριβώς η ΚΑΠ δεν είναι και τόσο μια πολιτική, δεν είναι και τόσο γεωργική γιατί ο δεύτερος πυλώνας είναι πιο σημαντικός και δεν είναι και τόσο κοινή διότι προχωράμε άρδιν στην επανεθνικοποίηση ορισμένων επιδοτήσεων. Τα πάντα τίθενται να αμφισβητήσει. Κοιτάξτε. Το θέμα αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Θα διατηρήσουμε το σύστημα των άμεσων πληρωμών σε αιτήσια βάση για κάποια περίοδο ή μήπως θα στοχεύσουμε μια συνελικότερη πολιτική στα πλαίσια της οποίας θα πληρώνουμε τους γεωργούς όταν υπάρχουν συγκυριακά προβλήματα και κρίσεις. Αλλά αν οι αγορές και οι τιμές είναι καλές, ο γεωργός δεν έχει κανένα δικαίωμα. Εμείς εξετάζουμε τις πολιτικές αυτές εδώ και αρκετό καιρό. Αν δείτε την αμερικανική εμπειρία, δεν είναι και πάρα πολύ καλή εδώ που τα λέμε, ούτε αυτή, ούτε σε επίπεδο κόστους αποτελεσματικότητας, ούτε και σε επίπεδο προβλεψιμότητας των δαπανών. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε ένα ετήσιο πλαίσιο δημοσιονομικό να έχουμε δέκα δις ας πούμε κόστος και το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 100 δις κόστος. Λόγω της συγκυρίας δεν γίνεται αυτό, θα δημιουργήσει διαρθρωτικά προβλήματα στον προϋπολογισμό. Μιλάμε για ένα θα έλεγα συμπαγές εξάντε καθορισμένο πολιετές δημοσιονομικό για έπτα αιτία που αγνοεί φυσικά τις κρίσεις και γι' αυτό ακριβώς δημιουργούνται όλα αυτά τα trust funds, τα υβριδικά μέσα. Έχουμε ξεφύγει πλήρως δηλαδή από το ετήσιο πλαίσιο. Λοιπόν θα δώσω τώρα το λόγο στον συνεισηγητή μας, τον μόνιμο συνεισηγητή, τον κύριο Ashworth ο οποίος θα βγάλει πλέον τα συμπεράσματα της ε, συζήτησης αυτής. Μιλήσαμε πολύ για την απλοποίηση. Υπάρχει η περιπλοκότητα που οφείλεται και στον πλούτο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την άλλη όμως τα κράτη-μέλη μπορούν να παρακάμψουν τις προβλέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και μιας και σε ορισμένες χώρες οι περιφέρειες έχουν πλέον την αρμοδιότητα να συνεισφέρουν και αυτές, έχουμε ένα τρίτο πλέον επίπεδο περιπλοκότητας να λάβουμε υπόψη. Όταν λοιπόν οι δικαιούχοι θυμώνουν εναντίον της περιπλοκότητας αυτής, είναι καιρός οι εμπλεκόμενοι να λένε κάθε φορά ότι φταίει η Ευρώπη. Κάτι το οποίο δεν αποδεικνύει δυστυχώς το ιδιαίτερο θάρρος το οποίο πρέπει να έχουν. Λοιπόν κύριε uh, Ashworth. Uh, Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Χόισλερ και να πω ότι αισθάνομαι και μια κατανόηση για την περίπτωσή του με τις όλες τεχνικές λεπτομέρειες που χρειάστηκε να μας δώσει και τις εξηγήσει, αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν πολύ, πολύτιμη η συμβολή σας. Από την πλευρά των τεχνικών λεπτομεριών, πολύτιμες πληροφορίες αυτές που μας δώσατε, εξηγώντα πώς λειτουργεί το σύστημα. Και Βεβαίω ε, η διαδικασία αυτή φώτισε κάποιες ιδιαίτερε πτυχές που πάντοτε μας απασχολούν. Ένα θέμα που επανέρχεται διακώ είναι η διακαής επιθυμία μας για απλούστευση. Το θέμα είναι πώς αυτό βέβαια θα εξισορροπηθεί ώστε να έχουμε την κατάλληλη αναλογία ε, από τη μια ευελιξίας και από την άλλη του κατάλληλου ελέγχου και λογοδοσίας. Και το πολιτικό στοιχείο που συζητήσαμε και με το οποίο ξεκινήσαμε ολόκληρο διάλογο είναι πώς οι διαδικασίε μπορούν να αλλάξουν ε, έχοντας υπόψη την ε, μελλοντική ΚΑΠ και πώς τα εργαλεία αυτά θα υλοποιούνται. Είμαστε στην αρχή όλης αυτής της συζήτησης, όμως ε, φωτίζεται η όλη προσπάθεια από τις σημερινές μας συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που μπήκατε στον κόπο να έρθετε και να συζητήσουμε. τιμη συνεισφορά. Να χειροκροτήσουμε τον κύριο Χόισλερ για τον χρόνο που μας αφιέρωσε, για τη σαφήνα των ε, ποντήσεων του και επειδή η τεχνική ε, είναι αυτός σκοπός, οι διαδικασίες είναι διαδικασίες, αλλά η πολιτική που είμαστε εμείς, η εκλεγμένη ε, πολιτική, επιβάλλει και η ΚΑΠ είναι ένα αντικείμενο που το βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της πολιτικής. Πρέπει λοιπόν πολλές φορές να αλλάζουμε τον προσανατολισμό μας ε, λόγω πολιτικών αιτίων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσέλευσή σας σήμερα. Συζητούμε για το ερχόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και νομίζω ότι έχουμε πλέον πολύτιμα στοιχεία στη διάθεσή μας για να εμπλουτίσουμε αυτή τη μεροντική εξέταση. Τώρα να δώσω το λόγο στους γενικούς μας εισηγητές, τον κύριο Γκέγερ για τον προπολογισμό 2017, τον κύριο Μουρεσάν για τον ε, επόμενο προπολογισμό 2018 και θα μας πούν για κάτι που είναι η μεγαλύτερη λαχτάρα των ε, ε, βουλευτών και που δείχνουν την προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε, τι γίνεται με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα δοκιμαστικά σχέδια σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά σχέδια, δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα μπορώ να σας μιλήσω για την προπαρασκευαστική προπαρασκευή ε, σχεδίων για το επόμενο, για το 2018. Όμως αυτό ε, θα το κάνει καλύτερα από μένα ο εισηγητή γι' αυτό το έτο. γιατί εγώ δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Yes, Mr. President, you are right. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν πιλωτικά προγράμματα και προσφατασκευαστικές δράσεις, ε, έχουμε διάφορα στάδια. Ε, θεσμία της 3ης Μαΐου ήταν ημερομηνία μέχρι την οποία μεμονωμένα βουλευτές, επιτροπές κτλ. έπρεπε στην Επιτροπή προπολογισμού να υποβάλουν τον κατάλογο πιλωτικών σχεδίων για να μπορέσει η Επιτροπή Προπολογισμού να στείλει ε, για πρόορη αξιολόγηση συγκομισιών. 344 στείλαμε για προ... προκατρακτική αξιολόγηση. Λάβαμε την αξιολόγηση της Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ θέλω να κάνω τώρα μία επισκόπηση. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει βαθμούς A, B, C, D στα project Α, A σημαίνει ότι μπορεί να υλοποιηθεί το πιλωτικό project όπως το προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 60 από τα 344 πήραν Α. Άρα η Κομισιόν λέει ότι αυτά μπορούν να γίνουν. 54 πήραν Β, B. Αυτό σημαίνει ότι εν μέρη μπορούν να υλοποιηθούν. Ή μπορεί και εξ ολοκλήρου εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει. Το Β, ο βαθμό Β σημαίνει ότι είναι καλό το πλωτικό πρόγραμμα, αλλά τελικά σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει προσαρμογή ή μερική προσαρμογή. Σύ πήραν πολλά 183 από το 344 που σημαίνει ότι αυτά τα οποία προτείνουν τα πιλωτικά προγράμματα καλύπτονται πλήρως από την υφιστάμενη νομοθεσία ή από νομοθεσία που έρχεται. Ή το θέμα καλύπτεται σε υφιστάμενα προγράμματα. Αυτό συμβαίνει συχνά να υπάρχει μια καλή ιδέα, αλλά να μην είναι γνωστό ότι αυτό καλύπτεται ήδη, χρηματοδοτείται ήδη από κάποιο υφιστάμενο πρόγραμμα. 47 τώρα πιλωτικά προγράμματα προπαρασκευαστικές ενέργειες πήραν το βαθμό ΔΕΛΤΑ, D, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή ότι είχαν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν, που σημαίνει ότι αυτομάτως ε, απορρίπτονται. Άρα, 60 πήραν α, πολύ καλά δηλαδή, τέλεια, 54 πήραν β, 183 σ και 47 δ. Και το είπα όταν επισκέφτηκα τις επιτροπές κοινοβουλευτικές. Είπα θα εστιάσουμε στα βαθμολογηθέντα με α και β project ε, που λέει η Επιτροπή ότι μπορούν είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρη να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν ή αν τέλο πάντων χρειάζονται κάποιες ελάσσονες αλλαγές. Όταν έχουν πάρει σε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα, σημαίνει ότι καλύπτονται από άλλου τομεί, άρα δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Και όταν έχουν πάρει το βαθμό δέλτα ούτε αυτά τα εξετάζουμε, αφού λέει η Κομισιόν δεν μπορούν να εφαρμοστούν, δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Άρα πήραμε την απόφαση να ε, εστιάσουμε στα α και β. 114 από 344 συνολικά project. Ένα τρίτο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε. Προπαρασκευασίε ενέργειε και πιλωτικά προγράμματα. Πόσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μα, να δούμε αν αρκούν και πώ θέλουν να προχωρήσουμε για τα πιλωτικά προγράμματα. Έχουμε 40 εκατομμύρια. Αυτό είναι το προβλεπόμενο ποσό. Για προπασκευαστικέ ενέργειε, για νέε προπαρασκευαστικέ ενέργειε, 50 εκατομμύρια είναι το ποσό συνολικά για προπαρασκευαστικέ ενέργειε, δηλαδή και για αυτέ που έχουν ξεκινήσει το προηγούμενο έτο, είναι 100 εκατομμύρια. Τώρα, το ποσό που έχουμε για πιλωτικά προγράμματα, όπω είπα, 40 εκατομμύρια. Αν δείτε τα πιλωτικά προγράμματα που πήραν Α, αν τα χρηματοδοτήσουμε 100% όπως ζητούν ε, τα μέλη, 46,9 είναι το σύνολο. Αν δούμε πλειοτικά προγράμματα που έχουν πάρει Α και Β, 105 εκατομμύρια είναι το ποσό, ενώ έχουμε 40 εκατομμύρια στη διάθεσή μας. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ λέω να κάνουμε το εξή. Θα ζητήσω από τις πολιτικές ομάδες, συντονιστές, σκιώδεις συζητητές, βλέπω κάποιους συναδέλφους εδώ παρόντες, και από το ΕΣΥΑΡ και από τους σοσιαλιστές. Σας παρακαλώ λοιπόν οι πολιτικές ομάδες να μου στείλουν μια λίστα προτεραιοτήτων. Τι θεωρούν πιο σημαντικό. Και θα τα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών Δηλαδή δεν θα χρηματοδοτήσουμε 15 προγράμματα από την Κούλτ και 0 από την ίτρια ή το ανάποδο. 15 από την ίτρια και κανένα από την Κούλτ. Πρέπει να ισορροπεί, Άρα θέλουμε να λάβουμε υπόψη τι πολιτικέ προτεραιότητε των ομάδων. Θέλουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των επιτροπών. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα αυτά τα καλά project που είναι καλά και τα α και τα β, θα ήθελα από αυτά τα καλά project να δρομολογήσουμε ώστε να το περισσότερα. Βλέποντας λοιπόν αυτά που είναι προτεραιότητα για τις πολιτικές ομάδες και για να έχουμε και ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών επιτροπών, αυτά τα δύο κριτήρια υπόψη, ε, είμαστε λίγο πιο πάνω από την οροφή, εγώ θα έλεγα να αυξήσουμε κατά 20-30% ε, τον προπολογισμό για να μην αφήσουμε πολλά προγράμματα εκτός. Δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα σωστά περισσότερα από αυτά καλά project να ξεκινήσουν. Αντί να συγγνώμη, όχι να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, να μειώσουμε λίγο αυτά τα κονδύλια που θα δώσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα ώστε να τον περισσότερα project και όχι να τα απορρίψουμε. Να μην κόψουμε δηλαδή το 20% αλλά ένα 30%. Θέλουμε λοιπόν όσο το δυνατόν περισσότερα project Α και Β να υλοποιηθούν, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε τι πολιτικέ σα προτεραιότητε για να δούμε τι μπορούμε να αφήσουμε εκτό και έπειτα να μειώσουμε τα ποσά για να μην βάλουμε σε κίνδυνο κάποια προγράμματα αν χρειαστεί να μειωθούν τα ποσά ή αν χρειαστεί να απορριφθούν κάποια project, μάλλον αυτό θα αφορά πιο πολύ τα B και όχι τα A. Όχι δηλαδή τα τέλεια, τα πιο καλά, για τα οποία δεν υπάρχει καμιά επιφύλαξη από την Κομισιόν. Αυτό θα προσπαθήσουμε να μην τα πειράξουμε. Για τις προπαρασκευαστικέ ενέργειες η κατάσταση είναι καλύτερη. Υπό ποια έννοια. Αν δούμε όλες τι προπαρασκευαστικέ ενέργειες, και να δούμε το Α και το Β που πήρανε και για τις ε, μάλλον την είναι για την άμυνα που προτείνει η Κομισιόν 106,6 εκατομμύρια. Και 100 εκατομμύρια είναι το ποσό. Άρα μικρή προσαρμογή θα χρειαστεί. Δηλαδή το προβλεπόμενο ποσό είναι 100 εκατομμύρια και αυτά τα project, αυτές οι προβλεπτικές ενέργειες θα κόστιζαν 106,6. Χρειαζόμαστε όμως, όπως είπα, τη συνεργασία των πολιτικών ομάδων και των επιτροπών. Αυτά, αγαπητέ Πρόεδρε, από τη δική μου πλευρά. Θα ήθελα λοιπόν τι επόμενε εβδομάδε να μου πούν οι συνάδελφοι τι θεωρούν σημαντικό. Θέλω επίση να πω ανοιχτά στου συναδέλφου το εξή. Τα πιλωτικά προγράμματα θα πρέπει να κατατεθούν ω δημοσιονομικέ τροπολογίε δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν έχουν υποβληθεί για προαξιολόγηση ότι έχουν ενταχθεί στον προπολογισμό. Το ξέρουν οι συνάδελφοι, αλλά μήπως και κάποιοι το έχουν ξεχάσει. Το επαναλαμβάνω για να τις καταθέσουν ως ε, τροπολίσεις του προπολογισμού. Αυτά είχα να πω και περιμένω τώρα τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων αλλά κυρίως ε, τη συνεισφορά των συναδέλφων τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. καταφέρατε πραγματικά να τα ε, χωρέσετε όλα σε αυτή την παρουσίαση, να κάνετε το αδύνατο. Μας προτείνατε, μας εξηγήσατε τις διαδικασίες, τι γίνεται με τις διαβουλεύσεις και τι μέθοδο μπορούμε να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ακολουθήσει αυτή την τόσο ορθολογιστική προσέγγιση. Ε, ίσως να θέλουν να παρέμβουν ο κύριος Δενανό και ο κύριος Βιώτη ή να θέσουν απορίες. Ναι, εγώ ήθελα να ε, παρέμβω για το θέμα αυτό. Είχα αναλάβει σε γιατί πριν δύο χρόνια. Ο διαγωνισμό που είχε ανακοινωθεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικέ ενέργειε ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτω οι προπαρασκευαστικέ ενέργειε θα λειτουργήσουν έτσι κι θα γίνει διαγωνισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη ερώτηση. Ίσως η Επιτροπή που είναι εδώ να μπορεί να απαντήσει. Ο κύριο Βιώτη. Ναι. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μούρεσαν, διότι πάντοτε είναι ακριβής, διεξοδικός και πειθαρχημένος στη δουλειά που αναλαμβάνει στα πλαίσια της κατάρτισης του προπολογισμού από δική μου πλευρά, από πλευράς, ε, πλευράς των σοσιαλιστών της ομάδας μας, θα υπάρξει στήριξη για την πορεία που προέγραψε ο εισηγητής και ως προς το μεθόδο εργασίας. Ως προς το πολιτικό περιεχόμενο προφανώς θα κάνουμε τη δική μας αποτίμηση που θα λάβει υπόψη τον τόπο, τι κατευθυντήριες γραμμές σε, κατά πρώτον τις κατευθυντήριες γραμμές στο Κοινοβουλίο τον, από τον περασμένο Μάρτιο, κατά δεύτερο λόγο την εντολή για τον τριμερή διάλογο που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ε, εδώ να ευχηθούμε για καλή τύχη, διότι θα αρχίσει να γίνεται από σήμερα, θα γίνουν από αυτή τη εβδομάδα οι πρώτε συναντήσει του τριμερού διαλόγου και μετά θα κάνουμε και μια πολιτική αποτίμηση στα επίπεδα τη ομάδα μα. Εκτιμώ ότι όταν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία πρέπει κανείς να κάνει τις κατάλληλες επιλογές. Δεν το λέω σαφώς ίσως και με αμεσότητα, διότι η μέθοδος εργασίας που θα υιοθετήσουμε δεν με πείθει πλήρως, δεν το λέω ειδικό, αλλά γενικώ. Δεν με ε, πείθει η προσέγγιση να προσπαθούμε να τους, να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Τέτοιες που λέμε στην Ιταλία, το να προσπαθήσουμε με ένα ε, κάλυμα να καλύψουμε τα πάντα δεν είναι εφικτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτεραιότητες, το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει συγκεκριμένε επιλογές, αρκετά συνεπείς, για να δώσουμε συγκεκριμένε αποκρίσεις στους πολίτες, ίσως με προγράμματα που έχουν ε, και ιδέες που έχουν προβάλλει κάποιοι συνάδελφοι. Υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές οι συνάδελφοι έχουν πει ποιε είναι οι προτιμήσει του. η συνεισφορά μα λοιπόν θα είναι προ αυτή την κατεύθυνση. Και σε μία ενθερμό αντίδραση για το έγγραφο, ε, όταν το λάβαμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαίνω ότι φέτο υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα ω προ την ε, κρίση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πιλωτικά προγράμματα που έχουν επιλεγεί. Δεν έχω τον αριθμό αναχείρας βέβαια, αλλά το λέω έτσι ως μια πρώτη αντίδραση με τη ματιά που έριξα. Ευχαριστώ. Αυτή η αυστηρότητα διευκολύνει τη δουλειά μας. Έχει κανείς άλλο σχόλιο, κύριε Όλμπριχτ. Δεν θέλετε. Πριν να ακούσουμε λοιπόν και πάλι το γενικό μας ασύγητη για να ολοκληρώσει, ποιος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα του κυρίου Ντενανό ένα πιλωτικό πρόγραμμα προδιετίας για το οποίο θα γινόταν ε, διαγωνισμός δεν έχει ε, γνωρίσει κανένα διαγωνισμό σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γενικό Εισηγητή για την πολύ καλή επισκόπηση. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε ευγνώμονες που ο εισηγητής σκοπεύει να περιορίσει την επιλογή των πιλωτικών προγραμματών και προπαρασκευαστικών δράσεων στις επιλογές Α και Β, όπως έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ε, ε, ήταν τεράστια δουλειά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις 344 προτάσεις και για μας είναι τεράστια ικανοποίηση. Το αποτέλεσμα αυτό, η προσπάθειά μας και ο καρπός του έργου μας λαμβάνεται υπόψη. Να σχολιάσω ίσως και το εξής. Σημειώνουμε την στρατηγική που διέγραψε ο κ. Μουρεσάν για να εκκινηθούν όσο πιο πολλά προγράμματα γίνεται και ή δυνατόν ή εφόσον δει μάλλον, να μειωθεί το ποσό ένα πρόγραμμα. Αυτό είναι εντελώ κατανοητό. Ωστόσο, εάν δούμε τη γενικότερη τάση που επικρατεί τα τελευταία δέκα χρόνια, βλέπουμε ότι η δυνατον η εφοσον δει να μειωθει το ποσο ενα προγραμμα αυτο ειναι εντελως κατανοητο ωστοσο οδηγεί σε σταδιακή μείωση του μέσου ποσού αναπρόγραμμα έτσι κι αλλιώ. Αυτό από μόνο του δεν είναι και καμία τραγωδία, όμως καλό είναι να το γνωρίζουμε. Εάν κοιτάξουμε το μέσο ποσό αναπληρωτικό πρόγραμμα, το 2009 ήταν 2 εκατομμύρια περίπου, ενώ το 2016, 2016 ε, την περσίνη χρονιά ήταν 250.000. Το μέσο ποσό για τις προπαρασκευαστικέ ήταν 1,5 εκατομμύρια το 2009 και αν δεν λάβουμε υπόψη και αυτές για τα ταμεία που τι στατιστικές, πέρσι θα ήμασταν μεταξύ του 1 και 1,5 εκατομμυρίου. Ένα γενικό σχόλιο για την τάση αυτή που παρατηρούμε και όσοι αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση για τις προπαρασκευαστικές δράσεις, για τις μέλησες θα πρέπει να το ελέγξω και να σας στείλω γραπτό στην απάντηση, διότι δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που θέτω την ερώτηση μου λένε θα σας απαντήσουμε γραπτός και ποτέ δεν έχω λάβει απάντηση. Θέλουμε απάντηση, αλλιώς θα θυμώσουμε. Έχετε βαριά ευθύνη, κυρία μου. Μέσα σε οκτώ μέρες πρέπει ο κύριος Ντελανό να λάβει απάντηση ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάψει να εγείρει υποψίες αδράνειας υπό αυτάς συνθήκας. Σε μία ε, εβδομάδα ε, θα είμαστε στην ε, πράσινη εβδομάδα και αυτό είναι καλό για τις μέλησες. Bon. Monsieur Κύριε Γενική Εισηγητά, για να ολοκληρώσετε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, ε, συμφωνώ και με όλου του υπόλοιπου, με αυτά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή πρέπει η δουλειά μα να έχει και κάποιο νόημα. Όταν λέω ότι θέλω να ξεκινήσουν ω το δυνατόν περισσότερα πιλωτικά προγράμματα και ε, για τα οποία είναι υπεύθυνοι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τρόπο, το είπα και προηγουμένω, να μειώσουμε το ποσό, αλλά όχι προβολικά, διότι η δουλειά δεν θα έχει κανένα νόημα ε, στην πράξη. Επίσης, και εγώ ίδιος είχα προτείνει πριν από δύο χρόνια ένα πιλωτικό πρόγραμμα και επόπτευσα την υλοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω ότι ο προπολογισμό είναι πολύ χαμηλός. Είναι απλώ πολύ δύσκολο να έχει ε, νόημα, να είναι λογικό ένα πιλωτικό πρόγραμμα, μια προσκευαστική δράση από μόνο του. Ε, τούτου λεχθέντος ε, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα προχωρήσουμε σε σοβαρέ περικοπέ για τα καλά πιλωτικά προγράμματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν έτσι κι αλλιώ. Και ναι, έχει δίκιο ο Ντανιέλα, διότι θα πρέπει να λάβουμε αποφάσει, να κάνουμε επιλογέ και να είναι σαφέ ότι οι πολιτικέ προτεραιότητε του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικές δράσεις. Οπότε, όπως είπα, θα προσπαθούμε να ε, επιλέξουμε τα καλύτερα που έχει ε, εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα α1β, αλλά να είστε βέβαιοι θα το κάνουμε με τρόπο ε, ορθολογιστικό και ε, να είμαστε σίγουροι ότι το κάθε πιλωτικό πρόγραμμα και αποπαρασκευαστική δράση που θα ξεκινήσει θα είναι προκοδοτημένο με αρκετό ποσό ώστε να έχει και νόημα στην υλοποίησή του. Αυτά από την πλευρά μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Merci, monsieur le rapporteur général. Ευχαριστώ, κύριε Γενική Εισηγητά. Ελπίζω την επόμενη φορά να συνυπογράψουμε όλοι ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, απλούστευσης των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Euh, Αυτό ήταν και μια παρότρινση για να πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο στο Γιάννης Γκέιερ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 2017 Αριθμός 3. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο δροτικού προπολογισμού υπαριθμών 3 που είναι λίγο πιο ασυνήθιστο σε σχέση με αυτό που γνωρίζουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το τρίτο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού προτείνει 500 εκατομμύρια ευρώ συμπληρωματικές πιστώσεις για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Αυτό να μπει στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, πληρωμές, έχουμε αρκετά χρήματα, αλλά για τις ανάληψεις υποχρεώσεων δεν είχαμε ε, ακόμη ξεκινήσει κάποιο κάτι στο τρέχον έτος, το συζητήσαμε διαμακρόν το θέμα. Και στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έκανε η Κομισιόν την πρόταση για συμπληρωματικές πιστώσεις ε, ανάληψων υποχρεώσεων 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση και καμία συζήτηση, γιατί το είχαμε ζητήσει. Αυτό που είναι λίγο περίεργο τώρα είναι ότι έρχονται και δύο προτάσεις ε, αλλαγής ε, σε ό,τι αφορά το οργανόγραμμα, τους πίνακες ε, δύο οργανώσεων, δύο οργανισμών, Άσερ και Σέζαρ 2. Αυτό είναι το περίεργο. επειδή μπορεί να προέρχονταν κάποια προβλήματα ή κάποιες απορίες, εγώ είδα ε, πάρα πολύ προσεκτικά ε, τις δύο αυτές προτάσεις ε, για τον Άσερ. Προτείνονται κάποιες ανακατατάξεις ε, στο, και σε προσωπικού, όμως ε, σε ό,τι αφορά το προϋπολογισμό δεν αλλάζει ο προϋπολογισμός του 2017, επομένως κατά την άποψή μου δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε αλλάζει και ο συνολικός αριθμός ε, των θέσεων και σε ό,τι αφορά το ΣΕΣΑΡ 2, που είναι μια κοινοπραξία. Εδώ έχουμε πάλι μια ανακατάταξη που αφορά τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή στην προκειμένη περίπτωση από άντε 14 να γίνει άντε 15. Είναι προσωποπαγής αυτή η ανακατάταξη. Επομένως, ε, επειδή θα λήξει ε, στο τέλος της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή, το δέχτηκε και το Συμβούλιο, τα προτείνει η Κομισιόν αυτά, δεν έχω εγώ αντίρρηση, δεν βρήκα κάποιο λόγο, επομένως, ε, παρότι είναι λίγο ασυνήθιστα αυτή η διαδικασία, προτείνω να δεχθούμε τις τρεις αυτές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τρίτο σχέδιο θεωρητικού προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γενικό Εισηγητή και παρακαλώ τους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να ε, πούν κάτι πάνω στην παρουσίαση από τον κύριο Γκάιερ. Θέλει κάποιος το λόγο? Από ό,τι φαίνεται καλύψατε τους πάντες κύριε Γενική Εισηγητά. Επομένως, σημειώνουμε αυτό που μας είπατε και περνάμε στο επόμενο θέμα, επιτροπή προπολογισμών. ή μάλλον για την ε, απόφασή μας 30 με 31 Αυγούστου θα καλυφθούμε να αποφασίσουμε στην Επιτροπή Υπολογισμών και ολομέλεια του Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν τροπολογίες που θα κατατεθούν προθεσμοί. Υπάρχει. Ναι, μια συγκινητική ημερομηνία 14 Ιουλίου για τη Γαλλία. 14 Ιουλίου λοιπόν προθεσμία εθνική γιορτή στη Γαλλία. Πότε, το μεσημέρι, α, στις 11, λίγη την ώρα που θα είναι η παρέλαση στα ηλίσια παιδεία δηλαδή. Eh Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λαβία για την πρόταση κινητοποίηση του Αλληλεγγύης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία που έζησε πολύ μεγάλα στις φυσικές καταστροφές με τραγικές συνέπειες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το Ταμείο Ελληνική για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδοτική βοήθεια για την Ιταλία, η οποία πραγματικά επλήγει σφοδρά από ε, μια σειρά σεισμών από τις 26 Αυγούστου 2016 έως τις 16 Ιανουαρίου 2017 ε, σεισμοί από τους 3,9 έως τους 5,6 σεισμούς της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε ε, πολλές περιοχές της κεντρικής Ιταλίας ε, το Λάτσιο, την Ούμπρια, τη Μάρκε και το Αμπρούτσο. Εδώ έπρεπε να δούμε την κινητοποίηση του Ταμείου για δεύτερη φορά το 2017 και επειδή ε, χρειάζεται να ε, κινητοποιηθεί 1,2 δις ευρώ ε, από τις μεγαλύτερες ε, από τα μεγαλύτερα ποσά που κινητοποιούνται για μιας. ιδίως για την περιοχή της Νόρτσα στην Ούμπρια. ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο των 229 ατόμων και περίπου 400 τραυματίες. Τον περασμένο Νοέμβριο ε, δεν είχαμε θύματα, όμως τον Γενάρη είχαμε άλλα 34. Χιλιάδες άνθρωποι ε, χρειάστηκε να εκενώσουν την περιοχή και όσοι χρειάζονταν βοήθεια ήταν περισσότερα από 30.000 κεφάλια στις τέσσερις περιοχές. Οι Ιταλικές αρχές υπολόγισαν το σύνολο των άμεσων ζημιών που φρούνται ε, στο σεισμό σε 2 δις ευρώ ένα ποσό που ξεπερνά το 1,3% του ΑΕΧ της Ιταλίας. Ως προς την κινητοποίηση του Ταμείου, αλληλεγγύης σε περίπτωση σοβαρών ζημιών είναι απαραίτητη παρέμβαση. Ε, είναι βαριά φυσική καταστροφή αυτή που γνωρίσαμε και για αυτό το λόγο το ποσό που προτείνεται είναι σκόπιμο συνολική διαθέσιμη πίστοση που ήταν στις αρχές του 2017 ήταν ένα δις. 563 εκατομμύρια ευρώ από το 2016 είναι χρήματα τα οποία δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν. Το ποσό τώρα αυτό λοιπόν για το 2017 φτάνει τα 902 εκατομμύρια ευρώ και 826. Αυτό ανταποκρίνεται στις συνολικές πιστώσεις της διαθέσιμες για το ταμείο, το, από πλευράς του Κοινωνικού Ταμείου είναι σαφές ότι με τα χρήματα του 16 τα οποία δεν έχουν καταναλωθεί και με συνολικά τα χρήματα του 17 δεν φτάνουμε το συνολικό ποσό και γι' αυτό θα είναι απαραίτητο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι να γίνει κάτι τέτοιο ε, και το επιτρέπει και το άρθρο 10 του κανονισμού του πολιετούς δημοσιονομικού έτσι ώστε τα χρήματα αυτά τα οποία πλησιάζουν το 1 δις να καλύψουν τις ανάγκες μέχρι το 2018. Απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού του 17 λοιπόν, ε, μια συμπληρωματική επιστολή λοιπόν, η υπαρίθμου 4 για το 17. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από αυτή το σκληρό χτύπημα ζητώ την υποστήριξή σας για την γρήγορη υιοθέτηση της ε, έκθεσης αυτής που θα επιτρέψει να αρχίσουν να δίδονται χρήματα αμέσω μετά το καλοκαίρι στην δύσκολη προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ιταλίας και βοήθειας προς αυτούς που τα πάντα έχασαν μετά από τον σεισμό. Ευχαριστώ κύριε Λαβία που υπενθυμίσατε τις τραγωδίες που χτύπησαν την Ιταλία και που ζητούν, απαιτούν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την εκδήλωση της ε, αλληλεγγύης. Το Κορεπέρ θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την πρόταση αυτή χωρίς τροπολογίες στις 12 Ιουλίου, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η υιοθέτηση της πρότασης αυτής, θα αποφασίσει το Συμβούλιο μέσω γραπτής διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να υιοθετήσει ε, στις 30 ή 31 Αυγούστου ε, την πρότασή της και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει κάποιος θέλει το λόγο. Α, ο κύριος Ντενανό. Όχι, εντάξει. Ο κύριος Ντενανό επιμένει. Εμείς υποστηρίζουμε την έκθεση Λαβία είναι απλό. είναι απαραίτητο, δεν μπορούμε να μην σταθούμε αλληλέγγυοι. Και εγώ, όπως και ο συνάδελφος Λαβία, ζητήσαμε να υποστηριχθεί πλήρως η προσπάθεια αυτή. 21 δις είναι οι άμεσες ζημίες, υπάρχουν και οι έμεσες ζημίες, τις έχετε διαπιστώσει και εσείς είναι περιοχές οι οποίες ε, οικονομικά, αν δεν υπάρξει αποκατάσταση οικονομική, καταδικασμένες σε θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καταστροφικές, ε, καταστροφικά συμβάντα θα πρέπει οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα γιατί η βοήθεια δίδεται τελικά πάνω από ένα χρόνο μετά τον δεύτερο σεισμό. 30 ε, εκατομμύρια προφανώς που δόθηκαν είναι σημαντικό ποσό, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά παρόλα αυτά οι ζημίες είναι πάρα πολύ υψηλές, τα ακούσατε και νομίζω ότι σε κατεπίγουσες καταστάσεις θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα και σε δημοσιονομικό επίπεδο να υπάρξει βοήθεια για την κάλυψη των αναγκών. Ευχαριστώ. Καλώς θα μείνουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα όπως είπαμε. Είπαμε η βοήθεια αυτή θα πρέπει να εγγραφεί στον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαρίθμων 4 για τον οποίο θα μας μιλήσει τώρα μόλις ο κύριος Γκάιερ. Ναι, αγαπητέ συνάδελφοι, έχουμε το σχέδιο Διορθωτικού Προϋπολογισμού υπαριθμών 4 για να εφαρμοστεί δημοσιονομικά και τεχνικά αυτό που στη, στην πράξη αυτό που μας παρουσίασε ο συνάδελφος Λαβία. Δεν θέλω να μακρύνω, τα ξέρουμε όλα τα γεγονότα. Πράγματι, πρόκειται για τις, ε, τη μεγαλύτερη συνεισφορά μέχρι τώρα από το Τάμιο Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το οποίο είναι κατανοητό λόγω του μεγέθους των φυσικών καταστροφών. Ζήτησε λοιπόν η Ιταλική κυβέρνηση περίπου 1,2 δις ευρώ, πολύ σημαντικό το ποσό αυτό, στο πλαίσιο και του συνόλου του προϋπολογισμού. Δεν αμφισβητεί κανείς ε, το λόγο, ε, τα είπαν και οι συνάδελφοι, καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαίο, αλλά 1,2 δις ε, δεν είναι και εύκολο να κινητοποιηθούν από τεχνικής πλευράς. Διότι μπορούν να εγγραφούν μόνο 500 εκατομμύρια και αυτό ουσιαστικά είναι εικονικό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή πρέπει να μεταφερθεί από άλλους τομείς. Και τώρα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο αυτό το ποσό. Και λέγεται στον δημοσιονικό οργανισμό ότι το 1 τέταρτο του ποσού δεν μπορεί να εκταμιευθεί μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Και το Συμβούλιο ε, ανησυχεί μήπως αδειάσει το ταμείο πολύ γρήγορα. Και μετά έρχονται και οι σεισμοί. Και αυτός ο φόβος γίνεται πραγματικότητα. Αυτό το οποίο προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά είναι ένας διπλός ελιγμός. Ήδη βάζουμε το χέρι μας και στον προπολογισμό του 2018 ε, με το λεγόμενο front loading, 300 εκατομμύρια. Και για τα υπόλοιπα που είναι απαραίτητα, λέει η Κομισιόν ότι μπορεί να διαθέσει αυτά τα κονδύλια από αυτά που είναι ήδη διαθέσιμα δηλαδή αν κατάλαβα καλά, από μη χρησιμοποιημένε πιστώσει από τα περιφερειακά προγράμματα για την περίοδο προγραμματισμού ε, μέχρι το 2013-2013. Τα είπαμε τα σχετικά με τον κύριο Χόισλερ. Αυτά που ήταν στα επιχειρησιακά προγράμματα της τελευταία περίοδου προγραμματισμού, εάν δεν έχουν ε, ε, χρησιμοποιηθεί κάποια κονδύλια, αυτά θα κινητοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Και θα ήθελα να μας επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι περί αυτού πρόκειται. Γιατί αν έχουμε την εκαθάριση των προγραμμάτων, αν όμως προκύψουν μετά και άλλοι λογαριασμοί, θα έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης και θα πρέπει να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για το προβλησμό του 2018 σε σχέση με αυτό που προβλέπουμε τώρα. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει αν αυτοί οι πρόσωποι που είναι εδώ σήμερα βέβαια μπορούν να μας ε, απαντήσουν. Αυτό που προτείνεται στο σχέδιο ε, διορθωτικού προϋπολογισμού 4, αν πράγματι μπορεί στην πράξη να ε, λειτουργήσει και να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά στενός κορσές αυτό ο προπολογισμό. Ευχαριστώ ε, που μας το, επιβεβαιώσατε και εσείς για μια ακόμη φορά. Αυτή λοιπόν η ακαμψία ε, δείχνει και ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη. Αδυνατή για ρυθμιστικούς, κανονιστικούς, νοσονομικούς λόγους ε, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αλληλεγγύης που νομίζω ότι όλοι το ε, καταλαβαίνουμε πόσο αιτιολογημένο είναι. Αν μπορεί λοιπόν να μας πει κάποια πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το κορσέ λοιπόν, ε, τον τόσο άκαμπτο, τον τόσο στενό, ε, πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτό το θεμητό αίτημα για τις φυσικές καθείς καταστροφές που ουσιαστικά έγινε το 2016. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το όντι. Νομίζω η συγητής πολύ καλά εξήγησε ήδη την δημοσιονομική δομή ως πιστώσεις για τον προπολογισμό το 2017 έχουμε 1,15 εκατομμύρια ε, δις ευρώ. Αυτό για το 2017. Αυτή ήταν ε, η μερίδα του 2017 και το 2016 εφόσον δεν είχε χρησιμοποιηθεί και βάσει του κανονισμού MFF. Αυτό το 1,15 δις δεν είναι 100% διαθέσιμο σε αυτή τη φάση της χρονιάς, καθότι, όπως είπε και ο εισηγητής, από το μερίδιο του 2017 το 25% πρέπει να παραμένει διαθέσιμο ως 1η Οκτωβρίου φέτος. 140 εκατομμύρια δηλαδή. Αυτά τα 140 εκατομμύρια δεν μπορούν να κινητοποιηθούν σε αυτή την φάση της απόφασης για τον σεισμό της Ιταλίας. Πρέπει να παραμένουν διαθέσιμο στο τέλος του τελευταίου τριμήνου της φετινής χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ε, ένα ποσό που λείπει. Κανονικά το ε, νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει σε έκτακτες περιστάσεις και φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούν εδώ ότι εδώ μιλάμε για πραγματικά ε, έκτακτες περιστάσεις να κάνουμε front loading να πάρουμε δηλαδή ένα κομμάτι από την τρανς, από την δόση του 2018. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να κάνουμε front-loading περίπου του μισού του ποσού της δόσης του 2018 για να φτάσουμε στο πλήρως ποσό του 1,8 δις. Αυτό σημαίνει ότι από το 18 θα πάρουμε 280 εκατομμύρια, ποσό μεγαλύτερο από την κατά μέσο όρο κινητοποίηση του Ταμείου ε, Αλληλεγγύης στη διάρκεια των ετών. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει λόγος να προδικάζουμε ότι αυτό δεν θα εξαρκεί, ιδίως εφόσον Μάλλον θα υπάρχουν κατά 140 εκατομμύρια που πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα για τι τελευταίου τρει μήνε τη φετινή χρονιά. Εάν δεν χρειαστούν ή χρειαστούν μόνο εν μέρη, και αυτά θα μεταφερθούν στο 2018 για να συμπληρώσουμε το ποσό των 280 εκατομμυρίων. Άρα, ελπίζω ότι διευκρίνησα την δημοσιονομική δομή που προτείνουμε και απλώς να επιβεβαιώσω ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουμε περαιτέρω αιτήματα υπό εξέταση. Βεβαίως όλοι θα γνωρίζετε ότι ένας σεισμός συνέβη πρόσφατα στην Ελλάδα και την Τουρκία μεταξύ των δύο χωρών και επίσης όλοι γνωρίζουμε τι καταστροφικές δασικές πρικαγιές είχαμε τον περασμένο μήνα στην Πορτογαλία. Έχουμε λοιπόν δύο ίσως μελλοντικές ε, αιτήσει στον αποτερορίζοντα θα τις απαιτημίσουμε εν καιρό, αλλά θα μπορούσαν εφόσον υποβληθούν φέτος να χρειαστούν μέρος των 140 εκατομμυρίων της φετινής χρονιάς και των 280 της ερχόμενης χρονιάς. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Γκάγερ για την χρηματοδότηση του ERDF, εάν μου επιτρέπετε, είναι εδώ ένα συνάδελφος της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο και να του δώσω τον λόγο για την ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα δεν είμαι ειδικό επί του προπολογισμού, αλλά πρέπει να πω ότι αληθεύει ότι τα κάτι μέλη πρέπει να έχουν αξιώσει ποσά για τα, προηγούμενα έτη προγραμματισμού έως τον Μάρτιο. Κάτι που δεν ε, συνέβη τελικά, ανάλογα με τα ποσά που διαθέτουμε, οπότε υπάρχει πλεόνασμα. Πλεόνασμα το οποίο μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αμέσως. Διατίθεται άρα. Για να μεταφερθεί για τους σκοπούς του Ταμείου Αλληλεγγύης. Μιλάτε για το ενδεχόμενο πλεονέσμα του έτους 2017. Μιλάτε για την ε, εκτίμηση για, προπολο... για στον προπολογισμό για το έτος 2017. Ναι, το όντι περί αυτού πρόκειται. Αυτό μου θυμίζει τη συζήτηση που είχαμε κάνει στα τέλη του 2014, όταν επρόκειτο να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονάσματα που είχαν προκύψει από έκτακτα έσοδα, πρόστιμα που είχαμε επιβάλλει σε πολυεθνικές εταιρείε που είχαν παραβεί το δίκαιο του ανταγωνισμού. Λοιπόν, ωραία. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να αποσπάσουμε Η ρευστότητα υπάρχει. Τα ποσά θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα. Ο κύριο ε, Όρμπικ θέλει να παραμπεί. Ναι, θα μιλήσω όμω στα πολωνικά γιατί είναι λίγο περίπλοκο το θέμα. Ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση στου εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να εξηγήσετε με κάθε ειλικρίνεια τι συμβαίνει με τα ποσά για την Ιταλία γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Θέλαμε να μετατοπίσουμε, να μεταφέρουμε κάποια ποσά από την ε, συνοχή. Αλλά είχαμε πει να μεταφέρουμε ποσά από τη συνοχή στην αλληλεγγύη για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Μα είχατε πει όμω τότε ότι οι διαδικασίε ε, του Ταμείου Λεγγύη είναι πολύ, πολύ χρονοβόρε. Γι' αυτό η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε προκατακτική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έλαβε και το Κοινοβούλιο στήριξε αυτή τη γραμμή με κάποιε αντιρρήσει. Άρα η Ιταλική κυβέρνηση έλαβε την έγκριση το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, ε, να αποδώσει ένα μέρος ε, των ποσών που διαθέτει από τη γραμμή για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Η Ιταλική κυβέρνηση όμως μας είπε τότε ότι ήθελε 200 εκατομμύρια ευρώ από το δικό της χαρτοφυλάκιο αμέσως. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τα πήραν αυτά τα ποσά εντός των Ταμείων Συνοχής. Από εκεί δηλαδή έγινε αυτή η μεταφορά. Διότι φαίνεται σαν να παίρνουμε χρήματα από τα Ταμεία Συνοχής και να τα πηγαίνουμε στο Ταμείο Λεγγύης. Δεν το πολύ καταλαβαίνω εγώ αυτό διαδικασία. Ήθελα κάποια διευκρίνηση, διότι είναι τα χρήματα της Ιταλίας, υπάρχει το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Λεγγύης. Πού βρισκόμαστε τώρα. Πού. Κοιτάξτε, είπαμε πριν στα πλαίσια της συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική ότι στην αρχή κάθε πολιετούς δημοσιονομικού προβλέπεται για κάθε κράτος μέλος μια σειρά πιστώσεων. Με μεγάλη ακρίβεια αυτό ισχύει και για τη συνοχή και για την ΚΑΠ. Α, και ο Σόλμπρεχτ λέει ότι προβλέπεται για την Ιταλία, το Ταμείο Συνοχής για την Ιταλία δεν χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ γιατί δεν θα μπορούσαμε προς το παρόν τουλάχιστον να πάρουμε από τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κύριε Πρόεδρε εμείς η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεχτήκαμε τη νέα διαδικασία η οποία νέα διαδικασία λέγει ότι η χώρα μέλος μπορεί να πάρει ένα τμήμα των πιστώσεων που προορίζονται γι' αυτό στο 100% λέει τώρα ο κύριος Όλμπριχτ και να ανταλλάξει ένα κομμάτι των χρημάτων αυτών χωρίς να υπάρξει συγχρηματοδότηση. Φεντέρ 100%, sans cofinancement. Λοιπόν, 100% ΦΕΝΤΕΡ χωρίς συγχρηματοδότηση το τμήμα το οποίο προβλέπεται για την περιφερειακή ανάπτυξη για την Ιταλία. Συμπληρωματικά η ερώτηση την οποία θέτω εγώ είναι αν θα μπορούσαμε στιγμιαία να χρησιμοποιήσουμε τις πιστώσεις αυτές και να τις επιστρέψουμε αργότερα όταν θα έχουμε μπορέσει να βρούμε στον προϋπολογισμό τα απαραίτητες πιστώσεις. Το θέμα είναι να θέσουμε το ταχύτερο δυνατόν στη διάθεση της Ιταλίας την ρευστότητα η οποία ανταποκρίνεται στην βοήθεια που θέλουμε να της δώσουμε. Ευχαριστώ. Να διευκρινίσω για την ερώτηση του κυρίου Όλμπριχτ. Δεν τίθεται θέμα να φύγουν χρήματα από τη συνοχή ε, στην αλληλεγγύη. Μιλάμε για δύο διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Από το Ταμείο Αλληλεγγύης προτείνεται μια κινητοποίηση 1,2 δις. Πέραν αυτού, συμπληρωματικά δηλαδή, υπάρχει μια συμφωνία έτσι ώστε να επιτρέψουμε με την συγχρηματοδότηση του 95% να υπάρξει συμπληρωματική χρηματοδότηση για την κάλυψη των ζημιών των σεισμών. Βέβαια τα συνολικά ποσά ε, εδώ φτάνουν οι ζημίες στο 20%. Το 5% θα πρέπει να προέλθει από το Περιφερειακό Ταμείο. Το 5%. Ένα δις δηλαδή περίπου. Στο εσωτερικό της Ιταλίας λοιπόν, τα χρήματα τα οποία δίδονται στις περιφέρειες θα μπορούσαν να αναπρογραμματιστούν εφόσον το επιθυμεί η Ιταλία για ένα ποσό μέχρι ένα δις. Ο κύριος Όλμπρεχτ μίλησε για 200 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Θεωρητικά λοιπόν η Ιταλία έχει το δικαίωμα να αναπρογραμματίσει τα ποσά αυτά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να στρέψει τα ποσά αυτά όχι στους αρχικούς τους προϋπολογισμούς αλλά στις περιφέρειες οι οποίες χτυπήθηκαν. Τώρα βλέπω τον συνάδελφο της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο, μην τυχόν θέλει το λόγο. Κοιτάξτε, έκανα λάθος. 95% όχι 100%. 95% για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, το διευκρινίζω. Κοιτάξτε, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε τώρα στο θέμα. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θέλει να σημειωθεί η εκκίνηση της διαδικασίας. Το ΚΟΡΕΠΕΡ θα δώσει την απόφασή του στις 12 Ιουλίου χωρίς τροπολόγηση για να υπάρξει επιτάχυνση της διαδικασίας αποδοχής του συμπληρωματικού. Θα υπάρξει συζήτηση γραπτά, θα υπάρξει απόφαση στις 4 Σεπτεμβρίου και εμείς στην συνάντησή μας στις 30 και 31 Αυγούστου θα τα συζητήσουμε και η ψηφοφορία θα γίνει στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι τροπολογίες στην έκθεση Γέγερ θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 14 Ιουλίου την 11η πρωινή. Ο κύριος Γκάιερ έχει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Όχι αλλά μια γενική ναι παρόλα αυτά. Νομίζω αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία διατίθεται το 2018 ε, στο Ταμείο Αλληλεγγύης ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πολύ βάσιμους λόγους, επειδή χρειάζεται η Ιταλία αυτά τα χρήματα. Το 2018 όμως το οικονομικό έτος δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και ήδη άδειασε κατά το ίμιση ο Κορβανάς για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Επομένως ε, θα πρέπει στις ε, ε, διαβουλεύσεις που θα έχουμε για το περιπλωσμό το 2018 να τα συζητήσουμε όλα αυτά γιατί μπορεί να υπάρξουν πλημμύρες, μπορεί να υπάρξουν σεισμοί, μπορεί να υπάρξουν άλλες φυσικές καταστροφές το 2018 και τα χρήματα τα οποία έχει το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα επαρκέσουν. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό με τους εταίρους μας ε, ε, για τον ε, προϋπολογισμό. Ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό πολιτικής πλευράς για μας. Πρέπει να το τονίσουμε. Ωραία. Έχουμε δηλαδή ενώπιον σε ένα πρόβλημα ασθένειας του προϋπολογισμού. Ο κύριος Όλμπριχτα, ίσως πρέπει να το πω τώρα αυτή τη στιγμή, ότι Υπάρχει και το αποθεματικό για τις φυσικές καταστροφές ε, που πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό, γιατί το σύστημα που έχουμε σήμερα δεν, απαιδεί, δεν αποδίδει, δεν λειτουργεί. Άρα πρέπει αυτό το αποθεματικό να το παλέψουμε να υπάρχει. Ναι, πράγματι. Θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη και δεν έχουμε τα εργαλεία, όπως διαπιστώνουμε. Άρα δίνουμε ένα θέαμα ανίσχυρης Ευρώπης στους πολίτες μας. Πρέπει λοιπόν ε, να φύγουμε από αυτό, για να μην δίνουμε ευρωσκεπτιστικά ε, επιχειρήματα. Η έκθεση του κ. Ντεπρέ, όπως είπα, να βάλετε για αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, όπω είπα, θα ξεκινήσουμε στις 9.30 και όχι στις 9. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αύριο το πρωί στις 9.30 επαναλαμβάνω με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εισηγητή τον κύριο Γκάιερ. Και θα ακολουθήσουμε με το θέμα του κυρίου Ντεπρέ. Δεν θέλει κανείς το λόγο. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι αύριο 9 το πρωί.